μέσα λοιπόν ad hoc, τα οποία του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και θέτουν το ζήτημα ε, ε, θέτουν κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να θέσουμε στην Κομισιόν σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των χωρών μελών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αυτά τα ταμεία. Δεύτερο ερώτημα είναι προκειμένου να πρικοδοτηθούν αυτά τα ad hoc μέσα. Χρησιμοποίησαμε πολλά άλλα μέσα όπως το μέσο της προένταξης, της γειτονίας, της συνεργασίας για την ανάπτυξη και τέλος φοβούμεθα ότι υπάρχει μια διάσταση μεταξύ των κανονικών ε, μέσων ε, στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Τώρα, όσον αφορά τον τίτλο 3, εδώ η κατάσταση είναι ακόμα πιο δεινή, ή ακόμα πιο δυσχερής θα λέγαμε ίσως, γιατί εδώ βρίσκουμε κάποια μέσα και διακυβέρματα που σχετίζονται με την κρίση του προσφυγικού όσον αφορά το Ταμείο χορήγησης, για τη χορήγηση ασύλου που είχε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από το 2003. Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας είχε μια αύξηση της τάξης του 15% σε πιστώσεις πληρωμών και εδώ βλέπουμε τις πιστώσεις για τα hot spots και η Frontex με μια αύξηση του, της τάξης του 98% για τις ε, υποχρεώσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η έκρηξη αυτή έχει τα ωριά της κάπου, δηλαδή έχοντας ε, ε, δεσμεύσει τα ανώτατα όρια, διερωτώμαστε τι θα γίνει στη συνέχεια. Και έχουμε πολλές ερωτήσεις σε σχέση με τις, τους δύο αυτού τίτλους, προσπαθώντας βεβαίω να παραμείνουμε στην διάσταση προπολογισμού έστω και έστω και αν πρόκειται εδώ για την πραγματικότητα αυτών των πολιτικών. Και θα έπρεπε να διευρύνουμε λίγο το θέμα, θέτοντας κάποια ερωτήματα εν σχέση με τη δυνατότητα δημοσιονομικής υλοποίησης αυτών των δράσεων, των επιγουσών δράσεων, για τις οποίες οι αποφάσεις λήφθησαν κατεπηγόντως γιατί υπάρχουν κάποιε αμφιβολίε εν σχέση με δυνατότητα υλοποίηση ορισμένων δράσεων, για παράδειγμα τα hot spots ή τα θέματα επανακατάσταση των προσφύγων. Άρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε στο τέλο ε, του χρόνου εν σχέση με την ε, χρήση αυτών των ε, πιστώσεων. Και βεβαίω θα υπάρξει μια σχετική συζήτηση μετά την παρουσίαση τη Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Τωμά. Νομίζω ότι το θέμα μας το παρουσιάσατε σαφέστατα. Η πολιτικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ δεν μα επιτρέπουν να ανταποκριθούμε σε τόσο σοβαρέ κρίσει όπω η μετανάστευση και πρέπει επίση να ανταποκριθούμε στην πραγματικότητα. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στην Τουρκία και διαπιστώσαμε ότι πέραν των ανακοινώσεων τα τρία δις από τη διευκόλυνση για την Τουρκία είχα, έχουν δοθεί μόνο 40 εκατομμύρια. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μεγάλες επιφυλάξεις ε, όσον αφορά των συνομιλητών μας και των ε, εταίρων μας. Κύριε Καρίνιο, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε Αρτουή, ευχαριστούμε κυρία Τομά για αυτή την εισαγωγή και σας ευχαριστώ για την συνεδρίαση αυτή, διότι πράγματι είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό και να δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά τη χρήση του κοινοτικού προϋπολογισμού και την απάντηση του κοινοτικού προπολογισμού στην πρόκληση της μεταναστευτικής κρίσης. Θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί ε, νιώθω πιο άνετα για την παρουσίαση. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι όλοι έχουμε την ίδια εντύπωση, την ίδια αίσθηση, ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει προκληθεί από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη γειτονία μας. Και έχει συνέπειες φυσικά σε θέματα ασφαλείας, σε θέματα κοινωνικών εντάσεων, έχει ανθρωπιστικές συνέπειες, πολιτικές συνέπειες και θεωρώ ότι όλοι ε, είμαστε και τρόπον την απογοητευμένοι. Το άκουσα και από εσά και συμφωνώ και εγώ, διότι θα θέλαμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε κατά τρόπον ώστε να ε, αντιμετωπίσουμε την κρίση με το πώς αποτελεσματικά θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως με το θετικό μήνυμα. Όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε καλό παράδειγμα ταχείας απάντησης από πλευράς των τριών θεσμικών οργάνων. Συνεργαστήκαμε προκειμένου να βρούμε όλε τις πιθανότητε μορφές ευελιξίε και όλου τους πιθανούς διαθέσιμου πόρους από κάθε γωνιά για να τους χρησιμοποιήσουμε εκεί που υπάρχουν οι ανάγκε. Και πράγματι, ε, χωρίς να αναφερθώ στο σεισμό στον οποίο αναφέρθηκε η κυρία Τομά, οι τίτλοι 3 και 4 ήταν σίγουρα αυτοί οι οποίοι ε, επλήγησαν περισσότερο από την κρίση και εγώ θα περιοριστώ στον τίτλο 4 γιατί ο τίτλος 3 είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί αργότερα εντός ημέρας. Να σας κάνω μια σύντομη ε, παρουσίαση των προϋπολογισμών που έχουμε, των πόρων που έχουμε διαθέσιμους και της κατάστασης στον τίτλο 4 με τα διάφορα ε, ταμεία που έχουμε και καταπιστεύματα που αναφέρετε στην εισαγωγή σας. Η πρώτη διαφάνεια δείχνει ένα σαφές παράδειγμα αυτού που σας έλεγα όσον αφορά την απάντηση από πλευράς προϋπολογισμού της Ένωσης το 2015-2016 έχουμε κινητοποιήσει περίπου 10 δις ευρώ για την αντιμετώπιση της ε, μεταναστευτικής κρίσης, διπλασιάζοντας τους πόρους που είχαν προβλεφθεί στον προπολογισμό. Και αυτό μας επιτρέπει φυσικά να επιβεβαιώσαμε ε, και αυτό που είπε ο πρόεδρος Αρτουή, ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν είχε ούτως ή άλλως προγραμματιστεί για να ανταποκριθεί σε αυτά τα ε, φαινόμενα κρίσης, τα ε, ποσά που είχαν προβλεφθεί ήταν ανεπαρκή, αλλά μπορέσαμε να διπλωσιάσουμε τα ποσά, διότι πέραν των 5,2 δις που είχαν προβλεφθεί από τα μέσα που ανέφερε η κυρία Τομά και στις εσωτερικές και στις εξωτερικές δράσεις, έχει ε, χρησιμοποιηθεί και ένα κονδύλιο 5,3 δις από τη χρήση ε, αποθεματικών στο τίτλο 3, στο τίτλο 4 και 1,8 δις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης που θα πήγαινε στο καταπίστευμα για την Αφρική για το διάστημα 2014-2020. Όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν χάρη πολύ σημαντικής ε, ε, επαναχρησιμοποίησης κονδυλίων, ε, χρήση του αποθεματικού κατεπίγουσας ανάγκης και το μέσο ευελιξίας που ξέρουμε ότι πολύ καλά από τους διαπραγμάτευση για τον ετήσιο προπολογισμό. Καταφέραμε λοιπόν να έχουμε ένα σημαντικό ποσό το οποίο θα είναι διαθέσιμο για τα όσα θα εφαρμοστούν στα πλαίσια αυτής της διετίας. Τώρα, ε, για να δούμε πώς επιμερίζονται τα διάφορα κονδύλια, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες ε, για τον τίτλο 3. Υπήρξε πολύ σημαντική ενέσχυση της κατεπίγουσες ε, βοήθειας στα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ενισχύσαμε επίσης τους αρμόδιους οργανισμούς, κυρίως το Frontex. Έχουμε δώσει κανδύλια στους ε, χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή και ένα ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα μετεγκατάστασης για τα άτομα που χρειάζονται προστασία. Όλα αυτά φυσικά δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε 15 μέρες, ούτε εν μία νυχτή, αλλά σταδιακά αρχίζουν και εφαρμόζονται. Όσον αφορά την εξωτερική μας δράση, νομίζω ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα εσωτερικά δεν θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί αλλού, Επομένω, πρέπει να επικεντρώσουμε τι προσπάθειε μα και στην εξωτερική δράση. Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε δύο δράσεις. Η μία αφορά τα πιο πιεστικά ανθρωπιστικά ζητήματα των προσφύγων και τι κοινότητές τους στις γειτονικές χώρες. Αναφέρατε και εσείς κύριε Αρτουή την Τουρκία, το Λίβανο, την Ιορδανία που είναι οι χώρε οι οποίες πιέζονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές. Επίσης, ε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη σταθερότητα και να αντιμετωπίσουμε ε, τα αίτια της παράνομης μετανάστευσης. Επομένως, δεν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τις ανάγκες των προσφύγων, αλλά να δώσουμε και κίνητρα στους ανθρώπους αυτούς να παραμείνουν εκεί που είναι. Το καταπίστευμα για την Αφρική είναι παράδειγμα αυτού. Πέραν του προπολογισμού προσπαθούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε όλες τις πιθανές πηγές μόχλευσης για τη βοήθεια για το ε, για τη μετανάστευση και μέσω της δημιουργίας των καταπιστευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω του μηχανισμού ε, για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Ε, η κυρία Τομάτα αποκάλεσε ad hoc μέσα, ναι μεν, αλλά δεν είναι απρόβλεπτα. Ο δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει τη σύσταση τέτοιων ταμείων, επομένως υπάρχει ένας προϋπολογισμός που είναι στη θέση να προβλέψει μέσα για μόχλευση και θεωρούμε ότι αυτό δεν θα συνεχίσει να είναι απολύτως ad hoc στο μέλλον αν θέλουμε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις. Τώρα, να περάσουμε απευθείας στον τίτλο 4. Τα τρία καταπιστεύματα που δημιουργήθηκαν, το καταπίστευμα για την Αφρική έχει προπολογισμό 1,8 δις για το 2016-2020, 405 εκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ένα πολύ σημαντικό κονδύλι είναι ε, συνεισφορά από το EDF και τα κράτη-μέλη έχουν συνεισφέρει ε, τα υπόλοιπα. <clears throat> Αυτά απαντά ένα από τα ερωτήματα που θέσατε, κυρία Τωμά καταπίστευμα Μαντάντ έχει λάβει 600 εκατομμύρια, 569 από τον ε, Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και 52 από τα κράτη-μέλη. Βλέπετε το συνολικό ε, ποσοστό που προέρχεται από τις διάφορες πηγές. Και για την διευκόλυνση για την Τουρκία, μετά από τις διαπραγματεύσεις, θα έχουμε μια πρικοδότηση 3 δισεκατομμυρίων, ένα τμήμα προβλέπεται για το 2016 και θα έχουμε και το αντίστοιχο ποσό στο σχέδιο ε, προϋπολογισμού για το 2017 και θα υπάρχει και ένα ποσό το οποίο θα δοθεί από τα κράτη-μέλη. Πέραν αυτών, όπως γνωρίζετε, ε, πριν από δύο εβδομάδες έγινε η διάσκεψη του Λονδίνου για τη Συρία, στην οποία τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκαν για ένα σύνολο τριών δισεκατομμυρίων. Το τμήμα του ευρωπαϊκού προλογισμού θα είναι 1,1 δις όπως επίσης και τη δυνατότητα μακροοικονομικής <laughs> ε, χρηματοοικής βοήθεια, που αν θυμάμαι καλά είναι 200 εκατομμύρια επιπλέον. Συνολικά αυτό σημαίνει ότι θα διπλασιάσουμε τη δέσμευση που είχε αναλυθεί στην προηγούμενη διάσκεψη. Τώρα, πέραν των τριών αυτών ε, καταπιστευμάτων, πριν αρχίσω να σας περιγράφω τα τρία καταπιστεύματα λίγο πιο αναλυτικά, η συνολική εικόνα του τίτλου 4 θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ε, ότι έχει ως εξής. Το 2016 ε, προβλέπονται 9 δις σε δεσμεύσεις, 2 δις σε πληρωμές, ε, που σημαίνει ότι έχουμε μία σε σχέση με πέρσι και επίσης να σας πω και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το γνωρίζω, είναι ότι χάρη στην καλή διαχείριση του προπολογισμού του 2015 και αυτό που προβλέπεται για το 2016, έχουμε καταφέρει να ε, διαγράψουμε τελείως τις καθυστερήσεις που είχαμε σε σχέση με την εκτέλεση των προηγούμενων προπολογισμών, που ήταν κάτι το οποίο θέλαμε οπωσδήποτε να, να περάσει ε, και να ε, βελτιωθεί στη διαχείριση. Επομένως, έχουμε βελτιώσει τις δεσμεύσεις μας στον τίτλο 4. Παρ' όλα αυτά, το 2016 ξεκινάει με μια ε, κατάσταση όπου έχουμε περιθώριο από θέματος 0 και έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά εκατομμύρια από το μέσο ευελιξία. Επομένω, το περιθώριο λιγμών που έχουμε στη διάθεσή μα είναι πάρα πολύ περιορισμένο για τον ε, τίτλο αυτό. Όπως σας επεσήμανα ήδη, το ευρωπαϊκά αυτά καταπιστεύματα είναι μέσα τα οποία μας επιτρέπουν να κινητοποιήσουμε τα κονδύλια ε, σε συνδυασμό με άλλους δωρητές. Τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, τα διάφορα προγράμματα τα οποία ε, υλοποιούνται βάσει του καταπιστεύματος έχουν νομική βάση και ακολουθούν τους κανόνες που έχουν εγκρίνει οι συνομοθέτες. Δεν παρακάμπτονται σε καμία περίπτωση οι κανόνες όσον αφορά την προενταξιακή βοήθεια και το μέσο ανάπτυξης και συνεργασίας. Ο Πρόεδρος, συγγνώμη που σας διακόπτω μισό λεπτό. για την ε, διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Υπάρχει συμφωνία για την κατανομή μεταξύ κρατών μελών, διότι δεν καταλάβαμε πολύ καλά αν τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να πληρώσουν τα δύο δις ε, τα οποία τους αναλογούν. Νομίζω πολύ εύστοχη ερώτησή σας, γιατί την τελευταία φορά που το συζητήσαμε ακόμα υπήρχε ένα κράτος μέλος που δεν είχε υπογράψει τη συμφωνία, αλλά πριν από δέκα μέρες ε, υπήρξε εν τέλει συμφωνία και όλες οι χώρες μέλη συμφωνούν να συνεισφέρουν και αρχίζουμε να ε, προετοιμάζουμε τον επιμερισμό των πληρωμών ε, ανάλογα με τις ανάγκες ρευστότητας ε, του καταπιστεύματος. Χαίρομαι που υπήρξε συμφωνία πριν από 10 μέρες. Μήπως όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενημερώθηκε. Συμφωνώ μαζί σας. Λυπάμαι που δεν σας ενημερώσαμε. Λείπαμε σε αποστολή την προηγούμενη εβδομάδα στην Τουρκία και δεν είχαμε την πληροφορία αυτή στη διάθεσή μας, ενώ η συμφωνία είχε ήδη υπογραφεί. Ε, θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ και να σας εκφράσω την επιθυμία να ε, επικοινωνούμε λίγο πιο σύντομα, ε, γιατί δεν είναι καλός τρόπος συνεργασίας αυτός. Έχετε δίκιο. Πράγματι, ήταν μια συμφωνία μεταξύ κρατών μελών, έγινε στο Συμβούλιο. Δεσμεύομαι να κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να σας ενημερώνουμε για τις ε, εξελίξεις. Ευτυχώς όμως πρόκειται για καλό νέο. Γιατί υπήρξε τελικά αυτή η συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και μπορούμε τελικά να προχωρήσουμε. Θα επανέλθω σε αυτό στο τέλος για να σας ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον μηχανισμό για την Τουρκία. Ήθελα επίση να τονίσω και να διασκεδάσω λίγο τις αμφιβολίε που υπάρχουν εδώ για τη λειτουργία των καταπιστευμάτων, λέγοντας ότι ε, αυτά τα ταμεία, ε, ε, τα προγράμματα που συμβάλλουν στα ταμεία υπόκειται σε κανόνες και εφαρμόζονται από την Κομισιόν, όπως προβλέπουν οι κανόνες. Και επίσης αυτά τα ταμεία υπόκειται στον ίδιο λογιστικό έλεγχο και εποπτεία και τις σχετικές προϋποθέσεις όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ε, κονδύλια. Οπότε από, αυτό το, αυτή την πλευρά υπάρχει το ίδιο σύστημα ελέγχου και εφαρμογής εκτέλεση των διαφόρων ε, κονδύλιων. Δεν θα μπω τώρα σε πολλές λεπτομέρειες με διάφορα, για τα διάφορα ε, ταμεία, γιατί οι συνάδελφοι από τις υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις θα σας αναφέρουν τα project που έχουν ξεκινήσει, οπότε να πάμε στην επόμενη διαφάνεια να τονίσω το εξής. Το Ταμείο Μαντάντ έχει ένα περιφερειακό πεδίο εφαρμογή, καλύπτει την Τουρκία, το Λίβανο και την ε, Ιορδανία, τα Δυτικά Βαλκάνια και το Ιράκ. Προς το παρόν έχουμε 390 εκατομμύρια τα οποία έχουν δεσμευθεί για να υπάρξει ε, στήριξη κυρίως στους τομείς της ε, εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της προστασίας παιδιών, καλύτερης πρόσβασης στην, ε, προς τις υπηρεσίες υγείας, σε βελτίωση των υποδομών νερού και απορριμμάτων και ανθεκτικότητα και οικονομικές δυνατότητες και κοινωνική συμπέριληψη. Οι συνάδελφοι θα σα δώσουν κάποιε πληροφορίε για το πώ ε, συνεχίζεται η εκτέλεση των ε, κονδύλιων αυτών. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα των project ε, αυτού του ταμείου που, που έχουν καταγραφεί εδώ στι διαφάνειε, αλλά θα αφήσω και πάλι του συναδέλφου να μπουν σε λεπτομέρειε. Τα οποία παραδείγματα όμως μας δείχνουν μια πολύ σαφή εικόνα για το τι περί πρόκειται και για το ότι όντως καλύπτουμε ή στοχεύουμε τις πραγματικέ ανάγκε όταν μιλούμε για την περιφέρεια αυτή και τις χώρες που βρίσκονται γύρω από τη Συρία. Το Trust Fund για την Αφρική τώρα είναι λίγο διαφορετικό, γιατί δεν επικεντρώνεται τόσο πολύ στην ανθρωπιστική πτυχή, αλλά έχει να κάνει με τις ε, βασικές αιτίες της ε, μετανάστευσης. Ε, ανθεκτικότητα, όπως είπα πριν, και δημιουργία υποδομών που θα βοηθήσει τους πολίτες να μείνουν εκεί που είναι και να μην θεωρήσουν ότι μόνη τους ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή είναι να μεταναστεύσουν. Υπάρχουν και σαφή παραδείγματα project στην Αιθιοπία ας πούμε Υπάρχουν διάφορα project για να βελτιωθεί η διατροφή, η επιστημιστική ασφάλεια. Στη Σομαλία υπάρχει η θελοντική επιστροφή των Σομαλών που βρίσκονται στην Κένια. Πάλι οι συνάδελφοι θα σα δώσουν περισσότερε λεπτομέρειε. Και να πω επίση ότι στι πρώτε συναντήσει τη Επιχειρησιακή Επιτροπή τα project ε, ύψου 101 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκαν για την ε, ε, περιοχή τη λίμνη Τσάτ και έχουμε ακόμα ένα σημαντικό ποσό που έχει δεσμευτεί για, την, για συνολικά για την, ε, περιοχή, για την Ήπειρο της Αφρικής. Τώρα, για τους ε, μετανάστες, για τους πρόσφυγες, συγγνώμη, στην Τουρκία. Όπω ξέρετε μέχρι τώρα υπάρχει ένα δισεκατομμύριο από τον Ευρωπαϊκό προπολογισμό και δύο δι από του προπολογισμού των κρατών μελών έχουν δεσμευθεί για τα έτη 2016-2017 στην Τουρκία. Είναι συντονιστικό μηχανισμό αυτό. θα έρθω σε αυτό σε ένα λεπτό. Τον διαχειρίζεται η Κομισιόν ω ε, κομμάτι του Ευρωπαϊκού ε, προπολογισμού. Υπάρχει, υπάρχουν αιτήσει εκθέσει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και υπάρχει πλήρη διαφάνεια και βεβαίω υπόκειται στι ε, αρχέ απαλλαγή. Ε, θα υποβληθεί η τελική εξέταση, ε, αξιολόγηση το 31 Δεκεμβρίου του 2019. Τώρα, τι γίνεται με τα τελευταία, τις τελευταίες εξελίξεις ε, για, την, για το μηχανισμό αυτό. Χτες, Είχα κάποιες, έλαβα κάποιες πολλές πολύ θετικέ πληροφορίες. Έγινε μια πρώτη διευθύνουσα, μια συντονιστική συνάντηση και υπήρξε μια σαφής αίσθηση ότι είναι επίγον το θέμα το σημαίνει ομόφωνη ε, απόφαση να αρχίσει άμεσα η εφαρμογή του τμήματος που αφορά τον, ε, το κομμάτι του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού για το 2016 επί τη βάση των αρχικών αναγκών και της αξιολόγησης που έγινε σε αυτή την φάση. Έγινε επίσης μία ε, διαβούλευση με τις τουρκικές αρχές και επίσης υπήρξε ομοφωνία για τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν κυρίως στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ανθρωπιστική πτυχή. Και επίσης τα project που υπήρχαν ήδη και είχαν ήδη δρομολογηθεί για την εκπαίδευση και για την, ε, για την κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών θα προωθηθούν ε, εν είδη προτεραιότητα στις επόμενες εβδομάδες. Και επίσης υπήρξε άλλη μια θετική εξέλιξη. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι θα, θα υπάρξει ένα συντονισμό των διαφόρων δράσεων των κρατών μελών στην περιοχή και θα υπάρξει μια χαρτογράφηση ώστε να υπάρξει αξιολόγηση ε, των συντονισμένων αυτών δράσεων. Αυτή λοιπόν η πτυχή της, ε, του συντονισμού του μηχανισμού αυτού της, ε, για την Τουρκία, για τους πρόσφυγες, ε, νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί. Κλείνοντας, να επαναλάβω αυτά που είπα στην αρχή. Θα θέλαμε όλοι η ανταπόκριση να είναι πιο ταχεία, να μπορούσαν άμεσα να υπάρξουν δράσεις επιτόπου, να μπορούσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε να λυθούν ή να έχουν ήδη λυθεί. Συμφωνώ, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό ακόμη, αλλά εντός του πλαισίου που έχουμε μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις πιθανές πηγές ευελιξίας για να μπορέσουμε να δώσουμε τους πόρους εκεί που χρειάζονται, εκεί που είναι οι προτεραιότητες. Τα παρατήματα 3 και 4 δίνουν, δείχνουν τους δύο βασικούς τομείς προτεραιότητας που είναι προτεραιότητα για όλους μας και νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί κομμάτι της βασικό τομέα της προσοχής μας και για το 2016 και σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Τομά στην εισαγωγική της παρέμβαση, το θέμα αυτό της ε, μετανάστευσης αλλά και όλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, που, προ, απορρέουν από την ε, οικονομική και κοινωνική κρίση, η κρίση ασφάλειας, νομίζω ότι θα αποτελέσουν τα σημεία που, στα οποία θα στοχεύσουμε στην ε, επόμενη, μέσα στην επόμενη χρονιά και σε αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε την απόλυτη προσοχή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καλβενιό. Επιτρέψατε μου να κάνω μια παρατήρηση όσον αφορά το μέσο διευκόλυνση για την Τουρκία γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τις χώρες μέλη. Η Επιτροπή ήταν τμήμα της κοινή συνεννόησης στη συνάντηση της 3ης Φεβρουαρίου με τις χώρες μέλη και η Επιτροπή βγήκε ε, στο να λάβει μία απόφαση. Το Κοινοβούλιο άρα θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά. Άρα η Επιτροπή ε, πράγματι έλαβε μία απόφαση ε, η κυρία Ζωζίαβα ε, είχε την πρόθεση να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και σε ποια προθεσμία και πρόκειται να διαβολευθεί επί της ουσίας το Κοινοβούλιο για την απόφαση αυτή. Ε, Κύριε Αρτουή, επιτρέψατε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι όπως το γνωρίζετε πολύ καλά είμαι απολύτως σύμφωνος ότι πρέπει να ενημερώνετε το Κοινοβούλιο και είμαστε απολύτως σύμφωνοι με αυτό. Ωστόσο, αναφέρεστε πιστεύω σε κάτι άλλο, το common understanding είναι μια συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών. Είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή επέτρεψε προσπαθώντας να καταλήξουν προς, μια, προς ένα common understanding και η Κομισιόν ε, ε, έλαβε αυτή την απόφαση ε, και εμπίπτει στη δική της αρμοδιότητα. Όσον αφορά για τον προπολογισμό, το Δεκέμβριο είχατε ενημερωθεί για τις ε, εξελίξεις ε, στο πλαίσιο των με τις χώρες μέλη και τότε θυμάμαι πολύ καλά ποια ήταν η συμβολή της Επιτροπής του προπολογισμού. Στην αρχή ήταν 5 εκατομμύρια, μετά 7 και καταλήξαμε στα 7 δις και αναφέραμε αυτά τα ποσά το Δεκέμβριο και δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε την ενημέρωση και θα κάνουμε μια δεδειγμένη πρόταση ε, όσον αφορά την κατάρτιση του προπολογισμού για το 2017. Θα υποβληθεί λοιπόν στην ε, φυσιολογική ετήσια διαπραγμάτευση και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμβάλλει ένα δις ε, μέχρι το 2007 για το μέσο διευκόλυνσης για την ε, Τουρκία. Υποθέτω ότι όλοι ε, πιστοποιούμε την ανάγκη να υπάρξει μια αναγκαία εισφορά εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Λυπούμε βεβαίως εάν έχετε την αίσθηση ότι δεν είχατε ενημερωθεί επαρκώς και θα προσπαθήσουμε να, είμαστε, να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο προσεχώς. Oui, merci, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Καλβινιό για όλες αυτές τις πληροφορίες. Ε, κατανοώ την απάντησή σας, αλλά όταν λέτε ότι αυτό αφορά το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ε, θα ήθελα να πω ότι παρόλα αυτά αυτό το μέσο διευκόλυνση για την Τουρκία δεσμεύει ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι κάπως, πώς να το πω, ε, ε, ε, με μια ευρία έννοια το πρόβλημα αυτών των θεσμικών οργάνων κατά την άποψή μου γιατί λέτε ότι τα ταμεία αυτά σχετίζονται με τα άλλα ταμεία, συναρτώνται με τα άλλα ταμεία, αλλά για ποια ταμεία πρόκειται εδώ. Πρόκειται κατ' ουσία για τη συμμετοχή των χωρών μελών ε, και του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελείται κατά 85% από τη συμμετοχή των χωρών μελών. Μόνο που στην πραγματικότητα έχουμε την εντύπωση πράγματι ότι πρόκειται για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος ε, τελικά χρησιμοποιείται με τρόπο ε, που υπεκφεύγει ε, των δημοκρατικών διαδικασιών. Και όλα αυτά δεν είναι... δεν εμφανίζουν καμία συνοχή και πραγματικά δεν υπόκειται σε κανένα είδου δημοκρατικού ελέγχου. Και διερωτώ με ποια είναι τα πραγματικά πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε μέσω της σύστασης νέων εργαλείων, νέων μέσων, γιατί εδώ υπάρχει μια απώλεια όσον αφορά την ορθολογικότητα ε, σε σχέση με τον ε, προϋπολογισμό, ε, την ορθολογική διαχείριση των ταμείων Έχω αμφιβολίες όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της σύστασης αυτών των μέσων που δεν είναι τίποτα άλλο παρά καινούρια μικρά κουτιά τα οποία, ε, ε, τα οποία δημιουργούνται κατ' ουσία με τη συμμετοχή των χωρών μολών. Και θεωρώ ότι οι κλέδες του επιμερισμού είναι λίγο διαφορετικές, παρόλα αυτά ε, προσωμιάζουν μεταξύ τους. Ευχαριστούμε κυρία Τομά. Μπορείτε να μας πείτε... Ε, ξέρω ότι έχετε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις, ε, κυρία Καλβίνη, οπότε θα πρέπει να φύγετε σε δύο λεπτά. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Τομά. Ναι, λυπούμε πάρα πολύ που πρέπει να φύγω, αλλά έχω μια υποχρέωση λιμένη αλλά ο κύριος Πρεσά και οι άλλοι συνάδελφοι θα παραμείνουν εδώ και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να αποκριθώ ε, στην κυρία Τομά. Η ερώτηση είναι εξή. Πρόκειται για μια βαλκανοποίηση του προπολογισμού, κατά την άποψή σας. Απάντηση, όχι. Δεν το πιστεύω και δεν το είχα πιστέψει πριν από δύο χρόνια όταν ξεκίνησα την εργασία μου στο, για τον προπολογισμό. Ε, ήταν ε, δεν πίστευα ότι ήταν ένα εργαλείο το οποίο θα αποκτούσε τόσο μεγάλη βαρύτητα. Ωστόσο υπάρχουν ε, πλεονεκτήματα ε, στη χρήση των καταπιστευμάτων και δεν βλέπω τα μειονεκτήματα τα οποία αναφέρεται. Καταρχήν μπορούν να κινητοποιηθούν κονδύλια πέραν από τα όρια του προπολογισμού και έστω και αν ε, έστω και αν υπάρχει μια σημαντική αύξηση του προπολογισμού, ε, θα προκύψουν καταστάσεις ενώπιον των οποίων ίσως δεν θα είναι αρκετοί οι πόροι. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα μέσο ε, κινητοποίησης των ε, πόρων και των κονδυλίων και μάλιστα αρκετά γρήγορα. Τα δύο δις για το μέσο διευκόλυνσης στην Τουρκία υπάρχουν, σε άλλα καταπιστεύματα υπάρχουν και η Νορβηγία και η Σουηδία που θα έχουν τη δική τους εισφορά. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν επιπλέον επιπρόσθετες δυνατότητες. Και αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο δεν έχουμε στο πλαίσιο του προπολογισμού αυτού καθ' αυτού. Δεύτερον, πρόκειται για τον ε, αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων. Και γιατί τον έφερα αυτό όσον αφορά το μέσο διευκόλυνση για την Τουρκία. Γιατί στην πρώτη συνάντηση υπήρξε ήδη μια ομόφωνη συμφωνία να υπάρχει συντονισμός ε, τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο σε επίπεδο των χωρών μελών. Και πραγματικά, ε, ειλικρινά, πρόκειται για ένα πολύ θετικό μέσο το οποίο πάει πέρα από τα όρια του προπολογισμού, ούτε ώστε η Ευρώπη να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και ε, θεωρώ ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τώρα, γιατί δεν θεωρώ ότι πρακτικά μια διαδικασία βαλκανοποίησης, γιατί το πρόγραμμα υφίσταται, τα προγράμματα υλοποιούνται, απλώς είναι διαφορετικό τρόπο να υλοποιηθούν. Ένας τρόπος που τελικά είναι πιο λογικός, γιατί πρόκειται για μια συνάρθρωση όλων των διακριτών μέσων και προγραμμάτων που έχουμε. Γιατί να έχουμε μια ανθρωπιστική δράση που να είναι εντελώς ανεξάρτητη από τις δράσεις για την ανάπτυξη. Είναι πολύ καλύτερα να υπάρχουν συνέργειες. Δηλαδή μια ανθρωπιστική δράση και μια ε, συνδυασμένη με μια περισσότερο ενβάθη δράση μέσω, για παράδειγμα, του εργαλείου ε, γειτονίας και των άλλων ε, δομών εξωτερικής δράσης. Το να έχει κανείς εργαλεία για το συντονισμό των διαφόρων μέσων, για να μην μιλάμε για το ΦΕΔ, ε, δεν πρόκειται για μια διαδικασία βαλκανοποίηση, αντιθέτω, πρόκειται για ένα πιο ευέλικτο τρόπο χρήσης των εργαλείων που έχουμε στο πλαίσιο του προπλογισμού, διασφαλίζοντας βεβαίω ότι διενεργούνται σωστά οι έλεγχοι έτσι όπως έχουν προβλεφθεί από τον συνομοθέτη και τελικά υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του ελεγκτικού οργάνου. Ε, Ευχαριστούμε, αλλά έχουμε εκλεγεί από τις χώρες μέλη και το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορεί ο, ο αυτός να είναι εύληπτος και να γίνει κατανοητός από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ένα θεσμός του οποίου ο προπολογισμός δεν είναι εύληπτος, κατανοητός από τον πολίτη ε, καθίσταται τροτός και ευάλωτος όσον αφορά ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Άρα λοιπόν, ε, λυπούμαστε πάρα πολύ που φεύγετε. Ο κύριος Περζάκ ε, θα παραστεί στη θα σας εκπροσπίσει στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους ε, για την παρουσίαση. Ευχαριστώ που αναφέρατε τις ανησυχίες σας για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020. Τα εργαλεία αυτά μάλλον εκπονήθηκαν πολύ αργά. Παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερως σημαντικά για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και εγώ αναρωτιέμαι αν ο τρέχον προϋπολογισμός είναι κατανοητός. Και ανησυχώ. Τι θα γίνει αν ξαφνικά χρειαστούν περισσότερα κονδύλια. Σε εργαλεία, σε ταμεία, τι θα γίνει αν τα κράτη-μέλη αρχίζουν να ζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη. Έχουμε να δώσουμε απάντηση εύλογη σε αυτά τα ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ταμείο για την Τουρκία, νομίζω ότι αναφέρατε 3 δισεκατομμύρια για το Ταμείο αυτό. Ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός θα συμβάλλει μισό εκατομμύριο και τα δυο, μισό δις, και τα 2,5 δις θα τα παράσχουν τα κράτη-μέλη. Αλλά τώρα έχουν ε, ε, επανεπολογιστεί αυτή, η, αυτά τα αριθμητικά στοιχεία και το 1 ε, δισεκατομμύριο θα παρασχεθεί από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εγώ θέλω να μου πείτε όμως το εξής. τι χρονοδιάγραμμα έχουμε, ένα μήνα, έξι μήνες, Έχετε ορίσει τη χρονική περίοδο μέσα στην οποία θα πρέπει να δοθούν αυτά τα κονδύλια. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ε, χρονικό όριο, το συντομότερο δυνατόν, για να μπορέσουν τα ταμεία Μαντάτ και Τουρκίας να λάβουν τα κονδύλια για να μπορέσουν να αρχίσουν να εφαρμόζουν όλες αυτές τις αποφάσεις και να, α, να εκτελούν τις διάφορες δράσεις. Επίσης, άλλο ένα ερώτημα. Έχουμε την δυνατότητα των εξοπλισμών να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα ταμεία αυτά εντός των Αφρικανικών χωρών και της Τουρκίας. Μπορούμε να ελέγξουμε όλα αυτά τα ad hoc εργαλεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριος Ντονανό. Ναι, ε, κύριε Πρόεδρε, προφανώς ε, συμμερίζομαι πολλές από τις απόψεις που εκφράσατε τόσο εσείς όσο και η κυρία Τομά. Εγώ αν κατάλαβα καλά η κυρία Καλβινιό μας είπε ότι αυτή η παράκαμψη του προπολογισμού θα οδηγήσει τελικά σε έναν αγκαίο συντονισμό. Ωστόσο, ε, θεωρώ ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Εδώ υπάρχει η δομική άρνηση των χωρών μελών να συμμετάσχουν σε αυτό το προεπολογισμό Και ε, εδώ γίνεται η προσπάθεια να παρακαμφθεί η βούληση των χωρών μελών. Ε, ε, εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη γενικά και η Κομισιόν ιδιαίτερα προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιες διαδικασίες που έχουν σαν αποτέλεσμα ε, να, να δημιουργήσουν κάποιες ε, αρνητικές ε, τελικά αντιδράσεις. Και φοβούμε ότι δεν θα είμαστε σε θέση σήμερα να υλοποιήσουμε αυτά τα ταμεία ή τα καταπιστεύματα είτε από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό είτε από τον προπολογισμό των χωρών μελών γιατί από πίσω υποκρύπτεται ένας απίστευτος εκβιασμός. Η πραγματικότητα βεβαίως είναι ότι θα πρέπει να παρεύουμε γρήγορα γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε απόγνωση που περιμένουν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ισχνά κονδύλια που φτάνουν και οι καθυστερήσεις μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θεωρώ ότι η Κομισιόν θα πρέπει σε σχέση με το προσφυγικό να εκπονήσει ε, κατεπίγουσες διαδικασίες και να ξεχάσει ίσως ε, όλες αυτές τις ε, καθυστερήσεις και το θέμα είναι να φτάσουν αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ο κύριος Δενανό έδωσε το κλειδί σε σχέση με τις αμφιβολίες αυτές γιατί εάν ακολουθούν οι ίδιοι κανόνες χρηματοδότησης ε, με όλες, όπως γίνεται συνήθως, γιατί τελικά ε, λέγεται ότι είναι ευέλικτα, ενώ δεν θα είναι. Ο συντονισμός ε, θα μπορούσε να γίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι, τέλος, ότι τελικά το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να δεχτεί έναν λογικό προϋπολογισμό όπως είναι αυτός ο οποίος επιθυμούμε και η Κομισιόν ε, προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια καταπιστεύματα εκτός του προϋπολογισμού ούτως ώστε να χρηματοδοτηθούν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί. Εγώ δεν λέω ότι δεν, έχουν, δεν έχει νόημα η χρηματοδότηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι παράλογο να πρέπει τα χρήματα αυτά να προέρχονται από τα μία και καταπιστεύματα εκτός του προϋπολογισμού. Και το πρόβλημα εδώ είναι το εξή. Πού βρίσκεται το Κοινοβούλιο, γιατί όταν είχαμε διαπραγματευτεί τον προϋπολογισμό για το 2016 ε, αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε για τον προϋπολογισμό. Η επικεφαλή των κυβερνήσεων ήταν στην ε, Λαβαλέτα. Ε, και η συμφωνία για τα τρία δις για την Τουρκία στη δική μας διαπράγματευση με το Συμβούλιο είχαμε προβλέψει μια αύξηση γιατί ξέραμε ότι θα τα χρειαστούμε για την ε, Τουρκία. Αλλά ε, τελικά ήταν άλλα τα ποσά τα οποία είχαν ε, προβλεφθεί τότε. Πού βρίσκεται λοιπόν το, το κοινοβούλιο. Τα δυόμιση θα και ποιος θα, θα, θα, πει όχι για όλα αυτά τα ποσά όταν τα ε, ποσά αυτά επιμεριστούν. Δεν νομίζω ότι κανείς ε, ε, θα αρνηθεί τα ποσά τα οποία είχαμε συμφωνήσει εμείς και δεν είναι τόσο πολύ μια καταγγελία που έχω κατά της Επιτροπής, αλλά πολύ περισσότερο ε, για τον ε, τρόπο που λειτουργεί τελικά το Συμβούλιο. Ε, το θέμα είναι ποια είναι η προστιθόμενη αξία εδώ. Ίσως δεν, χρειάζεται, δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά απαιτητικοί. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. θα πρέπει να σας πω ότι με τρομάζει η το ήρεμο πνεύμα των συζητήσεων, οι δηλώσεις ε, γεμάτες αυτοικανοποίηση εκ μέρους της Επιτροπής και η δυνότητα της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με έναν μικρό προϋπολογισμό, ενώ το ζητούμενο σήμερα είναι, το θέμα, το διακύβημα σήμερα είναι πόλεμος ή ειρήνη. Ε, αυτό το οποίο διακυβεύεται εδώ είναι το ίδιο το μέλλον της ε, ανθρωπότητας. Και αυτός ο ισχνός ε, προϋπολογισμός είναι ένας ισχνός προϋπολογισμός τον οποίον αποφασίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο οποίος δεν, ήταν, δεν είναι ενδεδειγμένος για να αντιμετωπίσει την κρίση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αφορά τον παράγοντα χρόνο. Δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στις κατεπίγουσες ανάγκες ε, κατασκευάζοντας ε, κάποια εργαλεία ενισχύοντας διαδικασίες ελέγχου. Είχαμε πάει σε μια αποστολή στην ε, Τουρκία και είδαμε σε ποιο βαθμό οι ίδιες οι δυσκολίες της ε, ε κινητοποίησης των ε, κονδυλίων τελικά έχουν σαν αποτέλεσμα ότι θα φτάσουν στους αποδέξεις τη στιγμή που έχει παρέλθει η κρίση. Και πραγματικά ε, τα καταπιστεύματα αυτά θα πρέπει να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Τελευταίο σημείο και αφορά το μελλοντικό προϋπολογισμό. Δεν βρισκόμαστε παρά στην αρχή της, αρχής του προσφυγικού προβλήματος και τελικά θα αναγκαστούμε να συνειδητοποιήσουμε σε ποιο βαθμό είμαστε παραπλησμένοι. Συζήτησα σχετικά με τον πρόεδρο κ. Αρτουή στην ε, Τουρκία, αλλά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό χωρίς να έχουμε κατά νου το ζήτημα των δημογραφικών ε, τάσεων ο παγκόσμιος πληθυσμός θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα είναι 12 ή 13 δις όταν η Αφρικανική Ήπειρος περάσει από 900 δις σε 400 δις. Πρόκειται για έναν τετραπλασιασμό ε, σκέψη η οποία θα έπρεπε να μας κινητοποιήσει γιατί αλλιώς θα βουλιάξουμε, ε, θα πνιγούμε στο πέλαγος των ε, ανεπαρκιών μας. Ευχαριστούμε ο κύριος Μαραγκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα το γεγονός ότι συζητάμε μετά από την εβδομάδα στην Τουρκία σημαίνει ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία πλέον διότι έχουμε το κεφάλι μας γεμάτο εντυπώσεις, εικόνες, ακόμα και συναισθήματα και πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο ψύχρεμοι εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Σίγουρα το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε μια σειρά, μάλλον είναι ενώπιον μια σειρά ε, τετελεσμένων. Και καλά κάνει ο πρόεδρος που το ε, διαπιστώνει και ε, υπερασπίζεται την νομιμοποίηση και την ανάγκη ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να έχουν το ρόλο που μας αναλογεί και που απαιτεί και η κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει και εμείς ως Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή να είμαστε διατεθειμένοι να εγκρίνουμε όλους αυτούς τους ε, μηχανισμούς ευελιξίας. Εάν υπάρχει ένας μηχανισμός συντονισμού μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών, τότε αυτή η ομάδα παρακολούθησης θα μπορούσε ίσως να βρίσκεται εδώ ε, και να είναι μαζί με το μηχανισμό συντονισμού, ε, ζώντας και δεχόμενοι τις αποφάσεις και βρίσκοντας ένα κατάλληλο μηχανισμό ε, για να εγκρίνει διαδικασίε απόφαση ή τουλάχιστον ακόμα και σε εσωτερικό επίπεδο εδώ στην Επιτροπή. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται και θα πρέπει να το ε, δεχτεί και αντιλαμβάνεται το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, μένα ε, δεν με ανησυχεί μόνο ο έλεγχος των οικονομικών αποφάσεων, αν είναι εντός ή εκτός του προπολογισμού. Με ανησυχεί και αυτή η εντύπωση που είχαμε και στην Τουρκία μιας κάποιας αταξίας, ε, αν όχι και χάος, ε, στην ε, αποτελεσματική εφαρμογή και στην πραγματική απόφαση του ποιος, πότε, για ποιο λόγο και πού θα εφαρμόσει αυτούς τους πόρους. Έχουμε το τράστ για την Αφρική, το μέσο διευκόλυνση για την Τουρκία, έχουμε τις ωραίες, έχουμε τα προγράμματα των κρατών μελών, έχουμε αυτά τα οποία συνεισφέρει η Τουρκία με όλο το θεσμικό της κόσμο. Έχουμε τα προενταξιακά μέσα, τα οποία υπήρχαν ήδη. Έχουμε 6-7, τουλάχιστον 6-7 πηγές. Εάν ε, δεν γίνει μια προσπάθεια να τα ε, πλαισιώσουμε όλα αυτά και να μπορέσουμε να τα παρακολουθήσουμε και να οργανώσουμε όλες αυτές τις πηγές χρηματοδότησης, ε, ελοχεύει ο κίνδυνος να χάσουμε κάθε έλεγχο για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, λαμβάνοντα δε υπόψη ότι πρόκειται και για μια κατάσταση ε, Δηλαδή, ε, σε σχέση με μια εβδομάδα πριν, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πραγματικά πόσος κόσμος είναι στην Τουρκία ε, και ποιοι είναι αυτοί οι υποθετικοί δύο εκατομμύρια άνθρωποι που δεν βρίσκονται στους καταβλισμούς. Υπάρχουν ε, και απτά προβλήματα, ε, παιδεία, στέγαση, προφανώς όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά είναι ένα μάλμα γαμά ε, ε, διέστησης και αυθόρμητης αντίδρασης. Και επίσης υπάρχει η απόδειξη στον προπολογισμό ότι έχουμε εξαντλήσει χρησιμοποιήσει τα περιθώρια, έχουμε χρησιμοποιήσει όλες τις ευελιξίες, αλλά δεν έχουμε εξαντλήσει το ενδεχόμενο να συμβούν περισσότερα πράγματα. Αν υπάρξει κι άλλη ε, ε, κρίση μπορεί να ε, δημιουργήσει πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει άλλη θα μπορούσε να ε, πολλαπλασιαστεί το πρόβλημα χωρίς λόγο. Ε, γι' αυτό νομίζω ότι και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δείξουμε δυνατότητα προσαρμογής και ε, να λάβουμε και αποφάσεις προφανώς. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητές μας λίγο πιο συντονισμένα και με πιο θετικό τρόπο, τουλάχιστον ακόμα και μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ε, η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία άλλωστε, λέει ο πρόεδρος. Η Ρωσία, η στάση της ε, ε, στη Συρία και στο Χαλέπι, οι απαιτήσει της Τουρκίας για τους Κούρδους στη Συρία, εχθές μία επίθεση στην Άγκυρα με αρκετούς νεκρούς και τραυματίες, η κατάσταση είναι ασταθής και πραγματικά χρειαζόμαστε και τα μέσα ευελιξίας. Καλύτερα να τα έχουμε αυτά εγγεγραμμένα στον προπολογισμό παρά να έχουμε προβλήματα χωρί να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ο λόγο στον κύριο Ντεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ακούω να μιλάτε, ακούω και τους συναδέλφου και σκέφτηκα τρία πράγματα. Πρώτον, νομίζω ότι μπαίνουμε σε νέα εποχή στο σχεδιασμό του προπολογισμού. Όταν ε, ακούμε τους ε, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, τρία πράγματα προκύπτουν συνεχώς. Πρώτον, μόχλευση, δεύτερον, προστιθέμενη αξία και τρίτον, προϋπολογισμός που να εκτελείται αποτελεσματικά. Και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αναρωτιόμαστε τι θα σημαίνει αυτό βαθμιδών και διαρθρωτικά στον προϋπολογισμό. Ε, δεύτερον, όταν διαπιστώνω με ποιο τρόπο λειτουργούμε, θα έλεγα, ε, όσον αφορά ε, εμάς ως Επιτροπή Προϋπολογισμού, ότι εμείς δεν είμαστε πια Επιτροπή Προϋπολογισμών και είμαστε απλώς ένα φορέας που κυρώνει αποφάσεις. Έχουν γίνει συζήσεις, συμβολογραφείο λέει ο Πρόεδρος. Μα ζητάτε απλώ να κυρώσουμε οι αποφάσεις, ε, στις οποίες ούτε ρωτηθήκαμε, ούτε και συμμετείχαμε. Ε, και πρέπει κάπως να ε, δοθεί μια κάποια νομιμότητα. Αλλά νομίζω ότι έχει μετατοπιστεί και το κέντρο βάρους των εξελίξεων. Ε, είδα εντάχει και θα συμφωνήσω με τα όσα ακούστηκαν μέχρι τούδε έκανα μια, ένα συσχετισμό μεταξύ των χρημάτων που θα προκύψουν από τα νέα τρία καταπιστεύματα τα οποία μας παρουσιάσατε και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι για τους επόμενους ε, χρόνους θα πρέπει να κινητοποιήσουμε 5,4 δις. Αυτό είναι το έγγραφο το οποίο θα μας παρουσιάσει ο κύριος Πρέζα. Εγώ το καλώ πιστώσεις Πρέζα ε, στον προπολογισμό, στον τίτλο 3, έχουμε κονδύλια για τη μεταμάστευση και είναι 3,8 για δύο χρόνια. Αν ερμηνεύω σωστά τις πίνακες που έχουμε εδώ ε, και μας δώσατε. Και νομίζω ότι θα υπάρχουν δύο ειδών συνέπειες ε, πέραν από τα ωραία λόγια. Εάν ζητούμε όλο ένα και περισσότερα από τα κράτη-μέλη να τροφοδοτήσουν αυτά τα, πιστεύματα, τους ζητάμε για το καταπίστευμα για την Αφρική, για το Μαντάτ και τώρα για ο μέσο διευκόλυνση για την Τουρκία. Θεωρείτε ότι θα έχουν δυνατότητα να δίνουν για τα ίδια πράγματα ε, τα ίδια ποσά και αυξημένα ποσά έχει ξεκινήσει ένας μηχανισμός όπου τα κράτη-μέλη θα τίνουν όλο ένα και περισσότερο συστηματικά να κλείνουν τη στρόφη του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιες πολιτικές. Σας το λέω ε, με ανησυχή, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη συνέπεια ότι σε αυτές τις ε, χρηματοοικονομικές προοπτικές, αν δείτε και τι προβλέπετε ε, για το μέσο διευκόλυνσης για την Τουρκία, οι κυβερνήσεις ξαναπαρεμβάνουν στα συντονιστικά όργανα. έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή για τον προπολογισμό, το οποίο κατά την άποψή μου ε, έχει συνέπειες τις οποίες μπορούμε να προβλέψουμε. Δεν χρειάζεται να προσπαθείτε εδώ να μας πείσετε ότι όλα αυτά είναι ανώδυνα. Ε, και συμφωνώ και με αυτά που έλεγε και ο κύριος ε, Μαζί προηγουμένως. Το πρόβλημα είναι ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδικασίας, διότι οι δημογραφικές τάσεις ε, δεν είναι τόσο αποκαλυπτικές όσο μας λέγεται. Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις ε, που σίγουρα θα επηρεάσουν ε, πάρα πολύ ε, τις ε, πολιτικές μας τα επόμενα χρόνια. Και λυπάμαι, αλλά αυτές οι πιστώσεις πρέζα πόρο απέχουν από τις πιστώσεις που χρειαζόμαστε. Ο κύριος Σάρβαμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας παρουσίασε το πώς έχει η κατάσταση. Δεν ε, μπορώ να πω βέβαια ότι είναι ένοχη για κάποιο έγκλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, αλλά ε, εν πάση περιπτώσει όχι ενσυνείδητα. Αλλά είναι πολύ λυπηρή η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ξέρω ότι όλοι εδώ στην αίθουσα συμμεριζόμαστε τους ίδιους στόχους. Ότι πρέπει όντως κάπως να διορθώσουμε την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν ε, ρομπότ πια και μπαίνει σε... Εδώ και χρόνια μάλλον ε, κινείται σε ε, σκοτεινά νερά Και πρέπει να πω ότι η καταιγίδα στην οποία βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή είναι προφανής. Είναι πολύ έντονη καταιγίδα η οποία χτυπάει τώρα το πλοίο μας, τη βάρκα μας και μάλλον θα κρατήσει και για πολύ καιρό. Είναι λοιπόν επίγουσα η ανάγκη να κάνουμε κάτι. Αυτό λοιπόν που συζητούμε εδώ τώρα είναι το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και η όλη δομή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και πώς αυτή πρέπει να αλλάξει αν τελικά θέλουμε να επιβιώσουμε από αυτή την καταιγίδα. Να επιβιώσουμε κυριολεκτικά, να μην βουλιάξουμε. Φοβούμαι λοιπόν ότι αυτό που σημαίνει όλο αυτό για την δομή του προπολογισμού είναι ότι θα, την, θα τον κάνει χίλια κομμάτια τον προπολογισμό μας και τώρα ε, επίτηδες είμαι τόσο δραματικός. Είμαστε το 2016 και έχουν αλλάξει τα πάντα από τότε που αποφασίσαμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν περιμένουμε μέχρι το 2019 2021 δεν θα είμαστε καν σε αυτή την αίθουσα πια κατά πάσα πιθανότητα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες επιλογές που παρουσιάζονται εδώ σε τούτο το έγγραφο και όντως έχουν χρειαστεί πολλή δουλειά για να υποβληθούν, αλλά δεν μπορούμε να διαλέξουμε κάποια από αυτές. Πρέπει να τις εφαρμόσουμε όλες ταυτόχρονα. Ο Ζεράρ είπε ότι είναι σαν ένα αυτοκόλλητο αυτό που βάζουμε εδώ. Τι θα μπορούσε να κάνει αυτό για να αλλάξει την κατάσταση. Θα αλλάξει τίποτα. Είναι κάποια πανάκια που μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα. Όχι. Είναι κάποιος επίδεσμος που βάζουμε πάνω στο πρόβλημα. Όχι. δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε απεργία. Τι να κάνουμε. Γιατί βεβαίως αυτό και αυτό θα είναι μια ε, κρίση που δεν είχαμε φανταστεί ότι θα εξελιχθεί έτσι, αλλά και η κρίση στην οποία βρισκόμαστε δεν είχαμε φανταστεί ότι θα εξελιχθεί έτσι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ένα μέρος της λήψης απόφασης, στα πλαίσια της συναπόφασης. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τον Πρόεδρο και όλα τα σχόλια που έκανε σχετικά με τη διαφάνεια κτλ. Αλλά για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ένα... όλα αυτά είναι έτσι ένα μικρό παρακλάδι του συνολικού προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο που ακολουθούμε λύνουμε τελικά το πρόβλημα. Βέβαια, όλα τα, τα πάντα καταλήγουν τελικά στο Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν έχουμε εκπρόσωπους του Συμβουλίου εδώ, αλλά τι γίνεται τελικά εκεί. Εγώ αν ήμουν ο Βλαντιμίρ Πούτιν, και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν είμαι, αλλά πραγματικά θα έκανα γιορτή κάθε μέρα, όλη μέρα. γιατί σε αυτό το χάος που επικρατεί στον κόσμο, αυτός είναι ο διευθυντής της ορχήστρας. Διευθύνει μια ορχήστρα εξαιρετικά και με την αδύναμη ηγεσία που είχαμε στη ΣΥΠΑ τα τελευταία 8 χρόνια, ας υπήρχε μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση να του αντισταθεί. Και αυτό φτάνει και στο Συμβούλιο, βεβαίως και σε όλα τα κρατη Ευχαριστώ grave que nous évoquons. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα που επικαλείστε, αλλά βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική κατάσταση και βλέπω ότι αγοράζουμε έπιπλα στο Πεκίνο ή στο Τόκιο για την 21η πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ίσως θα πρέπει να φροντίσουμε η διπλωματία μας και οι δυνατότητες άμυνας να είναι κοινέ, που το βασικό ερώτημα που τίθεται για το Συριακού κο είναι η ειρήνη και ίσως πράγματι ο Πούτιν να αποπειράται να ε, παίξει ένα παιχνίδι ανάμεσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία και την επιρροή του στη Σύρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με, τις, ε, με τους προηγούμενους ε, συναδέλφους. Να ευχαριστώ και εγώ την, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή του. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Πολύ σύντομα θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφος Ζαβαμά, αλλά και ο κύριος Ντεπρή. Είναι πραγματικά ε, έθεσε το δάχτυλο επί των τύπων των ήλων. Νομίζω ότι όντως εδώ ως ε, βουλευτές τούτου του Κοινοβουλίου θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο τι θέλουμε τελικά να επιτύχουμε. Και μια που σήμερα ακούσαμε πολλά ωραία λόγια, θα ήθελα να πω κι εγώ το εξής. Μου δημιουργείται η εντύπωση ότι εμείς είμαστε σαν, ε, σαν μια ομάδα γιατρών Αλλά υπάρχει και μια άλλη ομάδα γιατρών η οποία δεν μας έχει πει ποια θα είναι η θεραπεία της ασθένειας που διαπιστώσαμε ότι υπάρχει εμείς. Ξέρουμε ότι δίνουμε πολλά χρήματα, συμφωνούμε όλοι. Εγώ είμαι α, σύμφωνος με το να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά, αλλά δεν ξέρουμε τελικά ακριβώς πού πρέπει να πάει αυτή η βοήθεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει τελικά να φροντίσουμε εδώ όχι μόνο στην Επιτροπή Προπολογισμού, να συζητούμε για τα χρηματοπιστωτικά, τις χρηματοπιστωτικές πτυχές του θέματος, αλλά θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να, να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε τελικά με αυτό το πρόβλημα της μετανάστευσης. Εφόσον δεν ξέρουμε και κανείς από μας δεν ξέρει πόσα, πόσοι άνθρωποι θα έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Ε, πώς θα κάνουμε σωστό, πώς θα ε, χαράξουμε σωστή πολιτική για τον προπολογισμό αν δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι. Πού θα τους ε, ε, δώσουμε πρόσβαση αυτών των ανθρώπων ή στέγαση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα γενικό ε, πλάνο. Ό,τι και αν είναι το πλάνο αυτό. Θα πρέπει να είναι νομίμο, θα πρέπει, νομιμο, νομιμοποιημένο, θα πρέπει να είναι δημοκρατικό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Και προς το παρόν δεν, ε, δεν έχουμε καμία ιδέα για το τι θα γίνει. Ε, δίνουμε κάποια δισεκατομμύρια που από κάπου αλλού αποφασίζονται που θα πάνε και δεν ξέρουμε τελικά ποιος είναι ο τελικός μας στόχος. Πραγματικά κάνω έκκληση να αποφασίσουμε να κάνουμε μια σωστή, ένα σωστό προγραμματισμό γιατί τα κράτη-μέλη θα συναντηθούν και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσουν να συμφωνήσουν δυστυχώς για μια ενιαία λύση. Οπότε εμείς από εδώ πρέπει να ενισχύσουμε την χάραξη πολιτικής. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Φρυζά, αλλά και εγώ προσωπικά θα ήθελα να κάνω μιας... Ε, μερικές παρατηρήσεις, αν μου το επιτρέπει η Επιτροπή, η Κομισιόν. Είναι αλήθεια ότι η αποστολή μας στην Τουρκία μας εντυπωσίασε πολύ και είχαμε μια συνάντηση στο Τεπ με τον ε, υπεύθυνο της, ε, ε, της Ευρωπαϊκής, Κεντρικής Ευρωπαϊκής Μονάδας. Στην, στην, μας είπε ότι στην Τουρκία είναι μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων εκτοπισμένων και δεν μπορούν να φύγουν γιατί είναι κλειστά τα σύνορα και ότι αυτοί οι άνθρωποι οργανώνονται και βεβαίως κάποια μέρα ή άλλη θα προσπαθήσουν να διασχίσουν τα σύνορα για να μπουν στην Ευρώπη. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο αντιμετωπίζουμε δεν πρόκειται να σταματήσει. Και είναι αλήθεια ότι το πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι πραγματικά πολύ ευάλωτο και το να φύγει η Ελλάδα από το Σέγγεν γιατί δεν πληρεί σωστά τις υποχρεώσεις μου φαίνεται παράλογη γιατί στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα θα είχε ένα πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων από ό,τι σήμερα λοιπόν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι η λύση και έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δίνει εμφανίζεται εντελώ ανήμπορη και εφόσον βρισκόμαστε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, αντί να έχουμε αυτά τα πολλαπλά μέσα, αυτούς τους δεροφόρους γύρω από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό κάθε φορά μια επιτροπή διαχείρισης ε, για κάτι το οποίο θα έχει πολύ βαριές δικονομικές επιπτώσεις. Ε, ε, ε, δεν είναι δυνατόν οι πυροσβέστες να συζητούν που θα πάρουν το νερό. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε αυτή την εικόνα και δεν μπορούμε να συνεχίζουμε έτσι. Ε, πρόκειται για έκτακτους ε, πόρους στους οποίους χορηγούν τα κράτη επειδή η ενότητα του προπολογισμού είναι θεμελιώδης και αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει μια κρίση, υπάρχουν επιπρόσθετοι πόροι στον προπολογισμό που μπαίνουν. Δεν ε, πολλαπλασιάζονται τα διάφορα εργαλεία δορυφόροι γύρω από τον προπολογισμό έχουμε την αίσθηση ότι πειραματιζόμαστε συνεχώς ε, και δεν είναι, είναι εντελώ αδιαφανή ο προπολογισμό, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από κανέναν Ευρωπαίο πολίτη. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε σε κανέναν τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, προσπαθώντα εμβαλωματικά να καλύψουμε τι ανάγκε. Ε, και εγγράφονται στα έσοδα του προπολογισμού έτσι όπως προβλέπονται στο πολιετές δημοσιονομικό προπολογισμό όταν προστίθεται ένας τίτλος για έκτακτες ε, ε, καταστάσεις στην περίπτωση αυτή ο προπολογισμό έχει τις προβλεπόμενες ε, πιστώσεις και στη συνέχεια εφόσον υπάρχουν έκτακτες ε, συνθήκες γίνεται έκκληση προς τις χώρες ε, μέλη και λαμβάνονται από τον τίτλο 3 ή 4 τα αναγκαία κονδύλια χωρίς ε, να χρειάζεται να προστρέξουμε ακριβώς σε αυτά τα άλλα δορυφορικά εργαλεία τα οποία απογυμνώνουν το Κοινοβούλιο από τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου κύριος Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις, ξεκινώντας από μια διαπίστωση. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας ότι επίγει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της μετανάστευσης και το προσφυγικού με συντονισμένο τρόπο και να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις για την κρίση εντός και εκτός Ένωσης. Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχει μία τα, ε, ε, τάση να προσπαθήσουμε να δράσουμε ταχύτατα ε, και να επιτρέψουμε οι επιχειρησιακές αποφάσεις ε, να επιτρέψουν σε όλους τους φορείς να συμμετέχουν σε διαδικασία λήψης απόφασης με στόχο να αυξήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και παρκές έλεγχος για να γνωρίζουμε ότι τα κονδύλια των ε, εισφορών για τους πρόσφυγες ή τα ταμεία τα οποία θα δοθούν για την Τουρκία ή τα όσα θα προσθεθούν από τα κράτη-μέλη ε, στα καταπιστεύματα θα χρησιμοποιηθούν με σωστό, νόμιμο και ε, λογικό τρόπο. έχουμε λοιπόν αυτό κατά νου. Θα απαντήσω λίγο άτακτα στις ερωτήσεις. Τα καταπιστεύματα δεν είναι απαραίτητα μέσα τα οποία έρχονται να προσθεθούν, είναι μέσα τα οποία επιτρέπουν καλύτερο συντονισμό σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία πηγαίνουν πέραν των ορίων που καθορίζονται στη νομική βάση του κάθε μέσου που προκύπτει από τον προπολογισμό. Παραδείγματος χάρη, αν δούμε το καταπίστευμα για τη Συρία, το μαντάτ όπως το αποκαλούμε, που σημαίνει ελπίδα στα αραβικά, αυτό μας επιτρέπει να ε, έχουμε διάφορες πηγές προϋπολογισμού, τη γειτονία, την ένταξη, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ροής των μεταναστών, των προσφύγων μάλλον, που δεν είναι απαρατήτως ε, άνθρωποι που ε, θα μείνουν εντός ε, στενών γεωγραφικών ορίων ε, και μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο. Το Trust Fund μας επιτρέπει να απαντήσουμε ανάλογα με τις εξελίξεις και θα χρησιμοποιήσω και τον όρο που χρησιμοποίησε ο κύριος Σάρβαμα. Έχει καταιγίδα και η καταιγίδα μάλλον θα κρατήσει καιρό. Επομένως υπάρχει η ελπίδα της καλύτερης ε, συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών ε, που συνεισφέρουν ε, και κυρίως στους επόμενους μήνες θα φανεί αυτό στο Trust Fund. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να αυξήσουμε τα μέσα τα οποία διαθέτουμε και στην περίπτωση του μέσου διευκόλυνσης για την Τουρκία είχαμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε δύο δις ε, στα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα στον προπολογισμό και βεβαίως όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να επιστρέψω και στο θέμα ε, που ρωτήσατε κύριε Πρόεδρε για τη, ε, μέσω διευκόλυνσης για την Τουρκία και την ενημέρωση καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ώστε προκειμένου να μπορέσουμε να αποκρισταλώσουμε άποψη για την Τουρκία και να φτάσουμε στα 3 δισεκατομμύρια, χρειάστηκαν δύο μήνες από την ανακοίνωση σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων το Δεκέμβριο και της τελικής ε, συμφωνίας ε, στο Συμβούλιο, η οποία επιβεβαιώνει ε, ότι θα διατεθούν αυτά τα 2 δισεκατομμύρια που έρχονται να προσθεθούν στους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε και στην ανάγκη να έχουμε και κάτι, ένα τίτλο για τις έκτακτες περιστάσεις. Ε, ε, ίσως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προπολογισμό, αλλά όπως επεσήμανε και η κυρία Καλβίνιο στην παρέμβασή της, νομίζω ότι έχουμε αποδείξει συλλογικά ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα ευελιξίας που διαθέτουμε στον προπολογισμό ως Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα εδώ να προσθέσω και μέσω αυτών των καινοτόμων στοιχείων ε, το Trust Fund, αυτά τα, πιστεύματα και τους μηχανισμούς που προβλέπονται στο δημοσιονομικό κανονισμό. Υπάρχουν και κονδύλια εκτάκτου ανάγκης, τα οποία χρησιμοποιήσαμε και κάθε φορά ε, αποφασίζουμε για κινητοποίηση αυτών των ε, κονδυλίων του προπολογισμού. Ε, Επίση, η αρχή προπολογισμού μπορεί να χρησιμοποιήσει και το μέσο ευελιξίας, ε, κάτι το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στο έπακρο, ε, στον προπολογισμό του 2016. Προσπαθούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλα τα περιθώρια ελιγμών που διαθέτουμε. Για τον κύριο Μπερζέ που έλεγε ότι υπάρχουν προκλήσεις στην Αφρική, ο συγγνώμη, που ότι υπάρχουν προκλήσεις στην Αφρική. Αυτό το καταπίστευμα για την Αφρική ως στόχο έχει να επικεντρωθούμε σε κάποια από τα αίτια τα οποία αποτελούν και τη ρίζα των μεταναστευτικών ροών. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να επηρεάσουμε περισσότερο τα αίτια τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους να προσπαθήσουν να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον αλλού. Η χρήση λοιπόν αυτών των κονδυλίων και του Ταμείου Ανάπτυξης είναι ένας τρόπος να συνεισφέρουμε στην απάντηση, δεν είναι η πανάκια. Ο κύριος Μαραγκάλ ρώτησε πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα κονδύλια για την Τουρκία, για παράδειγμα, θα πάνε στους τομείς που απαιτείται περισσότερο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τις ανάγκες και η Διευθύνουσα Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ε, τα κράτη-μέλη και οι εκπρόσωποι ε, της Τουρκίας συμμετέχουν ως παρατηρητές προσπαθεί να διαπιστώσει ταχύτατα τι δράσεις απαιτούνται κατεπηγόντως. Και νομίζω ότι εκεί έχουμε προχωρήσει και προσπαθούμε να λαμβάνονται αποφάσεις ε, ταχύτατα ώστε ε, να εκταμιεύονται τα ποσά εγκαίρως, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατόν τις πιο επίγουσες καταστάσεις. Βέβαια, ε, εδώ υπάρχουν κάποιες εντάσεις και καταλαβαίνω και την απογοήτευση εδώ ε, δημιουργούνται εντάσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον προπολογισμό, αλλά θα έλεγα ότι ακόμα και για τον προπολογισμό του 2016 υπενθύμησε και κάποιος εδώ ότι στην τελική απόφαση στη ε, διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό το Κοινοβούλιο ήταν αυτό το οποίο κατάφερε να έχει την αύξηση στον προϋπολογισμό και χρειάστηκε αν επιπλέον κονδύλια και αυτά τα κονδύλια κυρίως για την Τουρκία ε, προσθέθηκαν στις ανάγκες και αυτό καλύπτει και το τμήμα το οποίο ε, έχουμε ήδη προβλέψει για το 2016. Υπάρχει ένα τμήμα για το οποίο ε, δεν είναι τόσο εύκολη η εκταμείευση. Θα πρέπει να περάσουμε από τον προϋπολογισμό ε, του 2017 ε, εξετάζουμε και τις πιθανότητες ε, χρησιμοποίηση άλλων κονδυλίων και αλλαγών ε, αν θεωρηθεί απαραίτητο. Άρα, νομίζω ότι από πλευράς δυνατοτήτων και ε, δράσεων μπορεί να μην αρκούν μένα, αλλά έχουμε. Όσον αφορά τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Ντεπρέ για τις προκλήσεις, αν αυτά δείχνουν μια τάση ε, τελείως διαφορετική σε θέματα προπολογισμού. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Αυτή η αίσθηση του κατεπήγοντος μας ε, ε, ε, εξωθεί να βρούμε όλα τα περιφέρεια ευελιξίας εντός και εκτός προϋπολογισμού ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. αν τα κράτη-μέλη τώρα είναι έτοιμα να διαθέσουν κονδύλια στον προπολογισμό της Ένωσης. Θα το δούμε στην ετήσια διαδικασία και φυσικά ε, θα το εξετάσουμε και στην ε, ενδιάμεση αναθεώρηση και θα δούμε κατά πόσον πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτά τα στοιχεία τα οποία συζητήσαμε σήμερα και να γίνουν οι πιθανές προσαρμογές ε, στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου όπως είναι καθορισμένο τώρα. Euh, Για να ολοκληρώσουμε, Νομίζω λοιπόν ότι έχουν υπάρξει δράσεις, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν διατεθεί. Τώρα αυτές οι εντάσεις επειδή ακριβώς επήγουν ε, κάποια πράγματα και υπάρχει και η διαδικασία λήψης απόφασης, υπάρχουν, υπάρχουν βέβαια ε, και προσπάθειες να ε, εκταμιεύονται τα κονδύλια όσο το δυνατόν πιο γρήγορα εκεί που απαιτούνται και πιστεύω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να κάνουμε και αιτήσεις, ε, συζητήσεις για τους ετήσιους προϋπολογισμούς του 2016, του 2017 και τα, στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης να προσπαθήσουμε λίγο να βρούμε από κοινού τις απαραίτητες λύσεις. Ευχαριστούμε κύριε Πρέζα να σας πω ότι και η κυρία Γεωργιέβο βα, πρέπει να περιμένει από μένα μια επιστολή διαμαρτυρίας για τον τίτλο 4. η ελληπής ενημέρωση της Επιτροπής Προϋπολογισμών μετά από τη συνεδρίωση της 7ης Φεβρουαρίου με τα κράτη-μέλη και ε, την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέπεια. Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα τις ε, συνέπειες ε, στο εσωτερικό ε, της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Ο κύριος Πρέζα θα λάβει το λόγο και πάλι και μετά ο Ματιές Σοέλ, ο οποίος είναι διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης HOME. 25 λεπτά αν μπορέσετε θα σας ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ και πάλι. Θα περάσω στα αγγλικά. Γιατί η παρουσίασή μου είναι στα αγγλικά. Θα προσπαθήσω να διατρέξω λίγο τις ε, διαφάνειες που επικεντρώνονται στι στις του προϋπολογισμού και θα αφήσω τον συνάδελφο Ματίας να μπει σε βάθος ε, για, τις, ε, για το πού βρίσκεται η εκτέλεση του προπολογισμού. Να ξεκινήσω αναφέροντας ε, κάποια βασικά οικονομικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις δαπάνες για την μετανάστευση στον τίτλο 3. Τα δύο χρόνια, τα δύο δημοσιονομικά έτη 2015 και 2016, τα μέσα που έχουν διατεθεί, να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, τα μέσα λοιπόν που έχουν διατεθεί για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ε, έχουν αυξηθεί κατά 80% για την ανταπόκριση στην, στις προκλήσεις της προσφυγικής κρίσης. Έχουμε πάνω από ένα 8 δις ευρώ, τα οποία έχουν προσθεθεί στις ε, διάφορες αποφάσεις, γραμμές του προπολογισμού, τροποποιώντας τον προπολογισμό και με την ε, τροποποίηση της σχετικής επιστολής. Ε, και ε, για την ατζέντα για την μετανάστευση, που ο στόχος της ήταν να συγκεράσει τις εθνικές προσπάθειες και τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σύμφωνα και με τις αρχές της μικτής ευθύνη και της επικουρικότητας, ε, το χρηματοοικονομικό πρόγραμμα που είχε προταθεί για τις ε, διάφορες υπηρεσίες μετακινήθηκε από τα 2,3 δις που είχαν ε, κατανομηθεί για τα τρία χρόνια αυτά και έφτασε τα 4,1 δις σε αυτά τα δύο χρόνια. Πού ενισχύσαμε τώρα τον προπολογισμό. Ε, σε ό,τι αφορά το μέγεθος, η μεγαλύτερη ε, αύξηση ήταν ε, στην συλλογική προσπάθεια για την επανεγκατάσταση. Πάνω από ένα δις δόθηκε για την επανεγκατάσταση των προσφύγων που υπήρχαν στην Ελλάδα και την Ιταλία. Επίσης υπήρξε μία ενίσχυση των δύο βασικών ταμείων του ασύλου και της μετανάστευσης και της ιστορικής ασφάλειας ε, με 310 ευρώ 310 εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη που είχαν χτυπηθεί πολύ έντονα από τη μεταναστευτική κρίση. Επίσης, υπήρξε τετραπλασιασμός των οικονομικών γραμμών για την επίγουσα βοήθεια. Ε, η ενίσχυση αυτή έφτασε τα 254 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Επίσης, σημαντική ενίσχυση της Frontex και θα ακούσουμε και από τον συνάδελφο από τη Frontex για το πώς οργανώνεται η ανταπόκριση από τη δική τους πλευρά. Συνολικά, στα δύο αυτά χρόνια, υπήρξε μία αύξηση 146 εκατομμυρίων ευρώ ε, για, την, ε, για τις επιχειρήσεις τρίτων και ποσειδών στην ε, Μεσόγειο, για, την, για τις επιστροφές και για την βοήθεια για την δημιουργία των hot spots. Επιπλέον, δόθηκαν 50 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης και επίσης ε, υπήρξε ενίσχυση σε ό,τι αφορά την, ε, τις ε, δυνατότητες ανταπόκρισης της Frontex και της Europol αλλά και της EASO σε ένα συνολικό, με συνολική αύξηση των, του προσωπικού με, σε, 143 επιπλέον θέσεις εργασίας. Πού είμαστε τώρα στο το 2016. Όπως υπόθηκε και πιο πριν, όλα τα στοιχεία της ευελιξίας ευελιξία έχουν χρησιμοποιηθεί για τον προϋπολογισμό του 2016 και το ε, περιθώριο δαπανών ε, και το περιθώριο ευελιξίας στο όριο δαπανών έχει χρησιμοποιηθεί. Το μέσο ευελιξίας επίσης έχει χρησιμοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε που σήμαινε και κινητοποίηση ε, περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Μηχανισμό Ευελιξίας για να αυξηθεί, ε, αυξηθούν οι δαπάνες για τον τίτλο 3. Στο 2016 λοιπόν, αν υπάρξουν επιπλέον ε, ανάγκες... Θα δούμε αν μπορούμε να ανακατανείμουμε τα ποσά μεταξύ του, του τίτλου 3, μεταξύ των προγραμμάτων του τίτλου 3, εάν δεν έχουν δαπανηθεί όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, αν αυτά δεν αρκούν, τότε ε, το τελευταίο μας μέσο ε, θα είναι να χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε το contingency margin για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα περιθώριο από τίτλους ε, σε, όλα το, σε όλους τους, ε, απογραμμές σε όλους τους τίτλους του προϋπολογισμού. Να δώσω τώρα το, τώρα το λόγο στον ε, συνάδελφο Ματίας για να σας πει για, τα, για τις λεπτομέρειες για την ε, εφαρμογή, για την εκτέλεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή που μου επιφυλάξατε σήμερα. Μέχρι τώρα ε, είχα, ε, ήμουν υπεύθυνο για την ε, πολιτική για το άσυλο, ήμουνα συνήθως προσεκλημένο από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, τώρα είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στη δική σα Επιτροπή. Θα ήθελα να χωρίσω την παρουσίασή μου σε δύο κομμάτια. Καταρχάς η κατάσταση σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των μέτρων για το 2015 και δεύτερον μια γενική έτσι, παρουσίαση της εικόνας για την ατζέντα για τη μετανάστευση και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το 2015 τα πρώτα, οι πρώτες συνέπειες των μέτρων που έχουν ληφθεί αρχίζουν να ε, υλοποιούνται. Επτά hot spots ε, είναι λειτουργικά. Ε, για την Ιταλία είναι το, η το Ποτζάλο και το Τραπάνι και στην Ελλάδα είναι στη Λέσβο, τη Χίο, τη Λέρο και τη Σάμο. να πω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η εκτέλεση του συστήματος ε, ε, μετεγκατάσταση πρέπει να ε, συνεχίσει την ε, πορεία της. Τα κράτη-μέλη έχουν, δεσμευτεί ότι θα μετεγκαταστήσουν 98.547 άτομα. Αυτό ακόμη πρέπει να εφαρμοστεί. Έχουμε 640 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν δεσμευτεί, δηλαδή 6.000 άτομα, 6.000 ευρώ συγγνώμη, για κάθε άτομο και 500 ευρώ για, κάθε, για, τα, για τα, ο κόστος μετακίνησης. Η εκτέλεση τώρα για τον, του μηχανισμού ε, μετεγκατάστασης ε, επίσης προχωράει καλά. Έχουμε περίπου 15.415 άτομα που θα μετεγκατασταθούν. Πάνω από 6.000 έχουν ήδη μετεγκατασταθεί. 153 εκατομμύρια ευρώ επίσης έχουν δεσμευθεί για το σκοπό αυτό. 10.000 δηλαδή ευρώ ανά ε, αξίωση και επίσης έχουμε 22.000 άτομα τα οποία θα μετακατασταθούν. Μπορεί αυτό να είναι χαμηλό, αλλά ο στόχος μας ήταν να έχουμε ένα πρόγραμμα πανευρωπαϊκό για τη μετακατάσταση και να μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα κρατημέλη, γιατί αυτό ήταν ιδιαίτερο σημαντικό θέμα από πολιτική πλευρά. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια Μέχρι τώρα έχουμε την, ε, τα, την ε, επίκουσα βοήθεια που δίνεται στα κράτη-μέλη στο σε ύψος 271 εκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια του Ταμείου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση για την προστασία της υποδοχής και την ε, διαπεξεργασία των αιτήσεων. Έχουμε 53 εκατομμύρια ευρώ που δεσμεύονται για την μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα. Από το 2015, από το Σεπτέμβριο του 2015, η Frontex έχει συντονίσει 16 πτήσεις και έχει ε, βοηθήσει την επιστροφή πάνω από 650 άτομα σε 6 διαφορετικές χώρες προέλευσης. Ο συνάδελφος από τη Frontex κατά πάσα πιθανότητα θα σας πει και άλλες λεπτομέρειες σχετικά. Τα εθνικά προγράμματα στα πλαίσια του ΆΜΙΦ περιλαμβάνουν 764 εκατομμύρια ευρώ που δεσμεύονται για την ε, ενσωμάτωση και, την, ε, και τα μέτρα για την νόμιμη μετανάστευση, καθώς επίσης και 605 εκατομμύρια ευρώ για επιστροφής. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασής μου, στην έβδομη διαφάνεια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να, είναι, να συνεχίσουν οι προσπάθειες ε, των κρατών μελών για να επιτευχθούν τα ορόσημα και οι στόχοι που έχουν τεθεί στα πλαίσια αυτής της μεταναστευτικής κρίσης. Μεταξύ μας νομίζω ότι ε, υπάρχει κοινή πεποίθηση σε ό,τι αφορά την, ε, τους στόχους μας, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Πέντε είναι οι βασικοί στόχοι που νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά την προσφυγική κρίση. Καταρχάς πρέπει να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Δεύτερον, πρέπει να αποκαταστήσουμε την πλήρη ελευθερία της διακίνησης εντός του χώρου Σέγγεν πέραν των τρέχουσών εξελίξεων που μας οδηγούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τρίτον, πρέπει να, έχουμε, να υποστηρίξουμε την, τα κράτη-μέλη εισόδου και αυτό σημαίνει δίκαιη κατανομή των προσφύγων μεταξύ των κρατών μελών και μια σταθεροποίηση καθώς επίσης και περαιτέρω ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Τέταρτος στόχος είναι η συνεπής επιστροφή των, ε, των απορριφθέντων ετούντων ασύλου και των ελαφρομεταναστών και πέμπτον η αντιμετώπιση των ε, γενεσιουργών αιτίων μετανάστευσης στην Αφρική και την Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε τώρα σε ό,τι αφορά την ε, δουλειά που γίνεται για να επιτευχθούν αυτοί οι πέντε πολιτικοί στόχοι. Τηλεγραφικά θα σας πω αναστόχο τι γίνεται και πού βρισκόμαστε. Στόχος 1 ασφάλεια στα εξωτερικά μας σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει το πακέτο για τα σύνορα τον Δεκέμβριο και όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις, ε, στη φάση των διαπραγματεύσεων, ε, περιλαμβάνει μια πρόταση για έναν εξ, ε, διευρυμένο ρόλο της Frontex για ελέγχους στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα. Επίσης περιλαμβάνει 7 νομοθετικές προτάσεις όπως αυτή για τα ταξιδιωτικά έγγραφα, για την, για την επιστροφή των παρανόμων διαμενών των μεταναστών και για την προσαρμογή του κώδικα Schengen. Συνολικά, περιλαμβάνει η πρόταση αυτή μια επιπλέον ε, δημοσιονομική προσπάθεια 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για να ενισχυθεί ο ρόλος του, της Frontex από το 2017 ως το 2020. Η πρόταση θα φέρει το, ε, τον αριθμό των ε, αξιωματούχων της Frontex στα 1000 άτομα το 2020. Πέραν αυτών, για τον πρώτο στόχο, να αναφερθώ και στο σχέδιο δράσης για την Τουρκία. Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν ε, να ε, ενισχύουν τις επιχειρήσεις ε, για, για τα 12 αυτά σημεία έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή του κοινού αυτού σχεδίου δράσης Ιδίω ό,τι αφορά τι εσωτερικέ πολιτικέ, ε, υπάρχει μια σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα εθελοντικό πρόγραμμα ανθρωπιστική υποδοχή, ε, το οποίο χάνει διαπραγμάτευση τώρα και ε, έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί, είχε προγραμματιστεί να συζητηθεί σήμερα με του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων και τον Πρωθυπουργό τη Τουρκία, ο οποίο δυστυχώ λόγω τη τρομοκρατικής επίθεση στην Άγκυρα ακύρωσε την επίσκεψή του. Έχουμε 80.000 άτομα εκτοπισμένα. Ε, και βεβαίως πρέπει να φροντίσουμε να καλυφθούν τα συγκεκριμένα κόστη που απορρώνουν από αυτό. Πάμε στους στόχους 2 και 3 που είναι η αποκατάσταση της Schengen ε, και η ε, σταθεροποίηση και η δίκαιη κατανομή των μεταναστών. Θα τους δω και τους δύο στόχους αυτούς από κοινού διότι συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Στον πυρήνα των συζητήσεων θα είναι ως προς αυτό τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες η μεταρρύθμιση του συστήματος Δουβλίνου. Οι βασικές προκλήσεις ε, που έχει το ε, σύστημα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να λειτουργήσει σωστά και οι, ώστε οι πρόσφυγες να κατανέμονται πιο δίκαια ε, και να αποφύγουμε δευτερογενείς μετακινήσεις. Παράλληλα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Δύο παραδείγματα θα σας πω έχουμε την ε, πρόθεση να εκπονήσουμε δείκτες ώστε να μπορούμε να ε, ελέγχουμε σε κάθε κράτος μέλος τα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να πληρούνται για τα κέντρα υποδοχής και επίσης μελετούμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε μια πρόταση για να υπάρξει ένα σύστημα αξιολόγησης για τις συνθήκες υποδοχής η οποία είναι, το οποίο σύστημα θα είναι παρόμοιο με αυτό της αξιολόγησης Schengen. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, τα δουλεύει όλα αυτά ταυτόχρονα. Από την οικονομική τώρα πλευρά του θέματος, η μεταρρύθμιση θα χρειαστεί περαιτέρω πόρους για να καλύψει τα κόστη μεταφοράς ε, της ε, διατήρησης των κέντρων υποδοχής και, την, και των υποδομών υποδοχής. Και θα καταλαβαίνετε βεβαίως ότι δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες εδώ, γιατί λόγω της πολιτικής κατάστασης δεν ξέρουμε ακόμα πού θα καταλήξουμε, πού θα, θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση από την σημερινή σύνοδο και από τη σύνοδο του Μαρτίου. Πάμε τώρα στον τέταρτο πολιτικό στόχο, συνολική ε, επιστροφή των ε, απορριφθέντων των ασύλων και, του, και των λαθρομεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ενεργός ε, στο να βελτιώσει την συνεργασία με το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, το Μαρόκο και την, ε, τις χώρες της Υποσαχαρίου Αφρικής. Και ο λόγο για τον οποίο επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα τρίτα κράτη για να έχουμε καλύτερε συμφωνίε συμφωνίες και καλώς λειτουργούσε συμφωνίε επανεισδοχή είναι ότι αυτέ οι χώρε είναι ε, χώρες ε, από τι οποίε έρχονται οι περισσότεροι μετανάστες ε, ε, πρόσφυγες στην Ιταλία και την Ελλάδα. να συνεργαζόμαστε και με την Frontex, τον IOM και άλλου, για να υπάρξει μια, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείριση επιστροφών και το πακέτο για τα σύνορα που σα ανέφερα ήδη του Δεκεμβρίου περιλαμβάνει προτάσει για να βελτιώσουμε βελτιώσουμε τη δυνατότητα που έχει η Frontex να υποστηρίζει την διαδικασία αυτή των επιστροφών. Ανεξάρτητα από τα όσα σας είπα ήδη, πρέπει να πω ότι ιδιαίτερος για, για το θέμα των επιστροφών, αλλά και για άλλους τομείς πολιτικής που σχετίζονται με το άσυλο και τη μετανάστευση, δεν έχουμε νομοθετικό πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα εφαρμογής το ποσοστό ε, επιστροφών ευρωπαϊκά ήταν 40% πέρσι. 60% ε, των ε, μεταναστών ή των προσφύγων που, δεν, που θα μπορούσαν να έχουν επιστραφεί δεν έχουν επιστρέψει στις χώρες τους. πέμπτος στόχος, αντιμετώπιση των γενοσυργών αιτιών για την μετανάστευση στην Αφρική και την Μέση Ανατολή. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί αυτό ξεπερνά την εντολή που έχει η Γενική Διεύθυνση Home οι δραστηριότητε αυτές ε, εμπίπτουν ε, στις εξωτερικές ε, πολιτικές κυρίω, αλλά να πω ότι στο δικό μας τον τομέα, τον οποίο καλύπτει η Γενική Διεύθυνση Home, εφαρμόζουμε την προγράμματα προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης με τη Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική και το κέρα τη Αφρική. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, να πω ότι το πλαίσιο στα οποία τα, τα, μία, τα, κονδύλια αυτά υποστηρίζουν τα κρατημέλη έχει αλλάξει, έχει τροποποιηθεί. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα, αλλά είναι μάλλον απρόβλεπτο και λόγω της, ε, ε, των ε, μεταναστευτικών ροών και των αναγκών που έχουν οι χώρες α, α προέλευσης, διαμετακόμισης και τελικές χώρες προορισμού ε, να δούμε, να, προς τα ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι ε, Ευρωπαίοι ηγέτες. Οι φάκελοι που σχετίζονται με τη μετανάστευση και που σας ανέφερα πιο πριν βρίσκονται στη φάση της διαπραγμάτευσης μερικώς. Ε, κάποιοι ακόμα συντάσσονται, οργανώνονται και μπορεί να αλλάξουν ε, το πολιτικό πεδίο και, τους, ε, και τα χρηματοοικονομικά μέσα. Με βάση μια απόφαση μπορεί να υπάρξει νέα πρόκληση η οποία μπορεί να είναι ότι τα κράτη-μέλη που δεν αντιμετώπισαν μέχρι τώρα την ε, προσφυγική κρίση όπως άλλα και που έχουν μικρότερη ε, δυνατότητα να κατανείμουν τους ε, πρόσφυγες θα έχουν μεγάλο μειονέκτημα γιατί η κατανομή των ε, κονδυλίων από την ΑΜΥΦ ε, ενισχύει κυρίως τις ε, χώρες που αντιμετωπίζουν στην πρώτη γραμμή αυτά τα προβλήματα της προσφυγικής κρίσης Ελλάδα, Ιταλία και άλλες. Και βεβαίως αφήνει σε δεύτερη μοίρα σε εισαγωγικά τις χώρες όπως οι βαλτικές χώρες που δεν αντιμετωπίζουν τόσο τραγικό πρόβλημα. Οπότε πρέπει να δούμε ποια θα είναι η πολιτική κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Πρέπει όμως να το έχουμε και αυτό υπόψη μας όταν μελετούμε τις μελλοντικέ οικονομικές ανάγκες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να διατηρήσουμε δυνατότητα που έχουμε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον ε, ε, μέσα ε, οικονομικά για τις συγκεκριμένες προτάσεις και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής πολιτική κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε εξαιρετικέ συνθήκε, ε, κύριε Πρόεδρε, το είπατε και εσεί, και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο χρειάζεται καταρχά ευελιξία στην εφαρμογή της ε, δυνατό, της, ε, των διαθεσίμων πιστώσεων που υπάρχουν. Είδα ότι και η δική σα επιτροπή έχει θέσει το θέμα αυτό ως στόχο της. Δεύτερον, Κατά πάσα πιθανότητα θα, χρειαστεί, θα χρειαστούν επιπλέον, ουσιαστικοί επιπλέον πόροι για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν στα πλαίσια του προπολογισμού 2017 και στην πρόθεσμη αναθεώρηση. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχετε εύκολο έργο και θα δούμε κατά πόσο οι επικεφαλής των κυβερνήσεων είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις ε, όσο δεν έχει λάβει χώρα το Βρετανικό δημοψήφισμα. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σακαρή Βερενσολά που είναι διευθυντής της, ε, ε, στη Frontex. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, επιτρέψατε μου επίσης να σας ευχαριστήσω πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω εδώ σε αυτή την επιτροπή και για μένα αυτή είναι η πρώτη φορά. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να ανταπεξέλθω στις προσδοσκίες σας. Δεύτερον, σας διαβιβάζω το μήνυμα από τον ε, εκτελεστικό μας διευθυντή, τον κύριο Φαμπρίτσιο Γκέρι, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και γι' αυτό εγώ τον αντικαθιστώ εδώ. Θα προσπαθήσω να διαφρώσω την ομιλία μου σε τρία τμήματα. Πρώτον, εν γενικά η κατάσταση στη Frontex. Δεύτερον, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στη Frontex και οι προκλήσεις και τρίτον οι μελλοντικέ προοπτικές και προκλήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν με, το, με τα πρώτα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση εν γέννη. Όπως συστήθηκε εδώ ήδη, αντιμετωπίζουμε ένα ευρύτερο φαινόμενο το οποίο αφορά τις αιτίες ε, εγκατάλειψης των ε, τρίτων χωρών όπου οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να αναζητήσουν προστασία. Ε, περνούν από χώρες διέλευσης, είναι στο έλεος των διακινητών και τελικά φτάνουν στο εξωτερικό σύνορο του Σέγγεν, της ζώνης Σέγγεν και εδώ αναλαμβάνει δράση Frontex. Και στη συνέχεια βρίσκονται και πάλι στα χέρια των αρχών των χωρών μελών είτε για χορήγηση ασύλου είτε για ένταξή του σε πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Άρα λοιπόν υπάρχουν, υπάρχει μια αλλαγή ε, στο σύνολο της εικόνας. Η Frontex είναι ο συνδετικός κρίκος της αλυσίδας στα εξωτερικά σύνορα. Προσπαθούμε να συνδράμουμε εκείνες τις χώρες που αντιμετωπίζουν ε, έκτακτη πίεση λόγω αυτής της κατάστασης. Και εδώ η Frontex είναι οργανισμός ο οποίος προσπαθεί να ε, χρησιμοποιήσει τα χρήματα τα οποία συζητάτε εδώ. Ε, αυτό είναι το ίμιση της λύσης. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι βεβαίως το πώς θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ούτω ώστε να βοηθηθούν οι χώρες οι οποίες υφίστανται αυτές τις πιέσεις. Και ιδιαίτερος σε αυτή την κατάσταση τώρα όπου η Frontex αυτή καθ' αυτή δεν έχει την εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή τα δικά μας στελέχη δεν επιτελούν αυτό το έργο είναι οι ακτοφυλακοί ιδιοκτικές αρχές των χωρών ε, μελών που έχουν την εκτελεστική εξουσία και εάν θέλετε κάνουν τη δουλειά. Η Frontex βρίσκεται εκεί για να διευκολύνει άλλες χώρες μέλη να πάνε να βοηθήσουν εκεί όπου παρίσταται ανάγκη τις χώρες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερους, τα μεγαλύτερα προβλήματα όπως είναι η Ιταλία και η Ελλάδα. Η Frontex λοιπόν βοηθάει τις άλλες χώρες να έρθουν να συνδράμουν, να υποστηρίξουν την Ελλάδα και την Ιταλία. Και εκεί πάνε τα περισσότερα από τα δικά μας, από τα περισσότερα από τα χρήματα, να, ούτε ώστε να χρηματοδοτηθούν ε, τα έκτακτα ε, στελέχη τα οποία συνδράμουν ε, την Ιταλία και την Ελλάδα επιτόπου στα hot spots ή όσον αφορά τη χρηματοδότηση επιπλέον περιπολικών, ελικοπτέρων ή αεροσκαφών για να ελέγχουν την περιοχή και να βοηθούν, ε, να υποστηρίζουν τον έλεγχο των συνόρων. Και βέβαια θα κατανοείτε ότι σε αυτή την κατάσταση όπου οι αριθμοί των προσφύγων που προσπαθούν παράνομα να περάσουν τα σύνορα έχει πραγματικά ξεφύγει, έχει εκραγεί. Ε, η Frontex δεν μπορεί να εξαρτάται ε, η Frontex εξαρτάται βεβαίως και από την ε, χρηματοδότηση. Αλλά όχι, δεν είναι δεν είναι το μόνο θέμα η επαρκής χρηματοδότηση, αλλά και η συνδρομή αυτή καθ' αυτή των χωρών μελών ε, που πρέπει να συνδράμουν με τους ε, δικούς τους ε, πόρους για να διευκολύνουν τις δράσεις μας. Αυτά όσον αφορά την γενική εικόνα. Πέρσι το 2015, όπως ακούσαμε, ο προπολογισμός μας είχε αυξηθεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από 114 δηλαδή σε 140 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, ε, αν το δούμε σε μια κλίμακα, είναι ε, μικρό το ποσό, αλλά για μας δεν είναι αμεληταίο. Και προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε την πρόσληψη περίπου 80 νέων ε, εργαζομένων στο προσωπικό μας και η πρόσληψη των στελεχών Α, συγγνώμη λέει ο ξέχασα να πω ότι παρόλο που έχουμε επιπρόσθετους ε, αξιωματούχους παρόλα αυτά χρειαζόμαστε περισσότερα στελέχη. Άρα η βασική γραμμή We συμμετείχε στις, στις ε, περικοπές κατά 5% του προσωπικού ε, παρόλο που χρειαζόμαστε περισσότερους. Ε, τώρα, η Frontex, ε, παρά τις προκλήσεις αυτές όσον αφορά τη μείωση του προσωπικού, η Frontex δεν είχε μια συμφωνία με την ε, Πολωνία. Αυτό σημαίνει ότι το καθεστώς μας στη χώρα αυτή, στην Πολωνία δηλαδή, είναι κάπως ασαφές και υπάρχει ένας μικρός ε, διορθωτικός συντελεστής για τις αποδοχές μας στην Πολωνία και όπως θα κατανοείτε η Πολωνία δεν είναι μέρος της ε, ζώνης ευρώ άρα υπάρχει υποκείμεθα στις ε, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η Frontex δεν είναι ε, ιδιαίτερα ελκυστικός ε, εργοδότης για τις παλαιότερες ε, χώρες μέλη. Αυτή ήταν μια πρόκληση ήδη το περασμένο χρόνο για μας. Επίσης η γλώσσα, το θέμα το γλωσσικό είναι ένα κάποιο πρόβλημα όταν υπάρχουν οικογένειες, σύζυγοι και παιδιά. Δεν είναι εύκολο να ενταχθούν στην ε, Πολωνία λόγω ακριβώς του γλωσσικού προβλήματος. Άρα τα περισσότερα στελέχη μας έχουν, ε, διαμένουν και στη χώρα προέλευσης και στην ε, Πολωνία. Τώρα, αν έρθουμε στο μέλλον, έχουμε σχεδιάσει το προπολογισμό για τα επόμενα έτη σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για το νέο κανονισμό για τη Frontex. Όπως ακούσαμε ένα στοιχείο του πακέτου της Κομισιόν είναι να δοθεί μια νέα εντολή προς τη Frontex, ένα, μια ευρύτερη εντολή και νέα καθήκοντα και ταυτόχρονα για τα επόμενα τρία χρόνια, το 17, 18 και 19, να αυξηθεί ο και να αυξηθούν και τα μέλη του προσωπικού μας. Άρα λοιπόν από τα 400 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, ο σκοπός είναι μέχρι το 2020 να πάμε στα 1000. Ε, και όπως είπα Όπω όπως εξήγησα ήδη, μπορείτε να φανταστείτε τι είδου ε, προκλήσεις ε, θα αντιμετωπίσουμε στο επίπεδο των προσλήψεων. Όχι μόνο λογιστικά προβλήματα, αλλά το πώς ε, θα βρεθούν 600 νέα εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία είναι ειδικευμένα ακριβώς στην, στο έργο των διοκτικών αρχών, ή στα, σε δραστηριότητες που αφορούν ε, την επαναπρόθεση των προσφύγων και τι αντίκτυπο θα έχει ε, στις ε, δυνατότητες των χωρών μελών να επιταλέσουν αυτές το ίδιο το δικό τους έργο. Άρα πράγματι θα έχουμε πολλές προκλήσεις στο μέλλον. Τώρα θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για το νέο, τα νέα καθήκοντα τα οποία σχεδιάζονται. Ήδη έχουμε δώσει στις χώρες μέλη αναλύσεις κινδύνου και συστάσεις όσον αφορά τους κινδύνους στα σύνορα. Και ήδη συντονίζουμε τις κοινέ επιχειρησιακές δραστηριότητε, ήδη ε, υποστηρίζουμε τις χώρες μέλη να επαναπροωθήσουν τους πρόσφυγες στις χώρες προέλευση, το κάνουμε ήδη. Η Επιτροπή προτείνει επιπλέον να αναπτύξουμε μια νέα λειτουργία ακτοφυλακής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των επαναπροθήσεων σημαντικά και αυτή τη στιγμή μέσω της Frontex ε, συντονίζουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες περίπου 3.000 ε, ε, περιπτώσεις ανά έτος αλλά μελλοντικά θα πρέπει ο αριθμός αυτός να δεκαπλασιαστεί. Άρα συνιστά μια μεγάλη πρόκληση για μας. Και επίσης θα έχουμε και άλλα καθήκοντα όσον αφορά την αξιολόγηση των αδυναμιών των χωρών μελών να επιτελέσουν το δικό τους έργο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μας και θα πρέπει εδώ να αναπτύξουμε το δυναμικό μας και τους πόρους μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω τυχόν ερωτή. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση μόνο. Η συμφωνία της έδρας έχει υπογραφεί με τις πολωνικές αρχές και τη Frontex. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι όχι, δεν υπάρχει συμφωνία με την έδρα, με την πολωνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ακόμα διαπραγματευόμαστε. Ε, η κυρία Τομά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δεν έχουμε πολύ χρόνο για τη συζήτηση, επομένως ε, θα πω απλώς ε, στον ε, εκπρόσωπο του Frontex ότι συμφωνούμε και εμείς με τις δύο βασικές σας ανησυχίες, την ευελιξία δεδομένου ότι είναι δύσκολο να προβλέψουμε επακριβώς στην κάθε λεπτομέρεια πιάστε στις εκατοντάδες των ευρώ που θα χρειαστούν και επίσης να πω ότι ε, πρέπει να υπάρξει και αναπροσαρμογή που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες που πόρα απέχει από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είδαμε ότι ο προπολογισμό του 2016 χρησιμοποιούσε πολύ περισσότερα πόσα είχαμε στη διάθεσή μας, ε, περισσότερα από το παρόν περιθώριο ευελιξίας και πραγματικά θα ήθελα να έχω μια εικόνα για το πώς, για το πώς ε, θα ε, διαμορφωθεί το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Διευθυντά και για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ανοσυχώ ακόμα περισσότερο μετά από αυτά που μας είδατε, από ό,τι ανησυχούσα πριν, ε, διότι μας αναλύσατε και τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν όσον αφορά την έδρα, το καθεστώς, ε, την απουσία ανθρώπων που να θέλουν να έρθουν να εργαστούν, αυτό νομίζω ότι ε, αποκαλύπτει ε, πόσο επίγοντα είναι τα πράγματα. Επομένως, ε, μας ενδιαφέρει μεν ο συντονισμός των ε, υπηρεσιών, αλλά χρειάζονται και συντονιστές για να κάνουν συντονισμό των υπαλλήλων. Και δεν ξέρω τώρα όσον αφορά το θέμα αυτό, ίσως δεν κατάλαβα καλά για τον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι αναφερθήκατε σε ένα δις. Ε, για την ακτοφυλακή. Ε, τι να σας πω, για αυτό τον προϋπολογισμό προς το παρόν ακόμα, εκτός και αν μου διέφυγε εμένα, δεν ε, ξέρουμε από πού θα το πάρουμε πάλι, τι αλλαγή θα κάνουμε. Ε, τι να σας πω, ένα νέο μέσο ε, επιπλέον προπολογισμού της Ένωσης ε, για να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όλο ένα χάος είναι. Να σας καθησυχάσω κυρία Τομά, έχουμε ακόμα 35 λεπτά για τη συζήτηση. Μείνετε ήσυχοι. Ίσως θα μπορούσατε και εσείς να ρωτήσετε πού θα είναι αυτοί οι χίλιοι, ποιοι θα είναι στη Βαρσοβία και πού θα είναι οι υπόλοιποι. Κύριε Διευθυντά, μήπω θέλετε να απαντήσετε στην κυρία Τομά και στη συνέχεια ε, δεν ξέρω ποιο θέλει να λάβει το λόγο, μπορεί να λάβει το λόγο. Καταρχά όμω να απαντήσετε στην κυρία Τομά. Monsieur le Président, Κύριε Πρόεδρε, προσπαθούμε να συντονιστούμε λίγο ποιος θα απαντήσει τι. Λοιπόν, να απαντήσω καταρχάς στην ερώτηση της κυρίας Τομά για τις συνέπειες για τον προπολογισμό, για την δημιουργία της υπηρεσίας ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής. Πρόκειται για ένα κονδύλιο μέχρι το 2020, επομένως υπάρχει προγραμματισμός ε, στον τίτλο 3 ο οποίος αυξάνεται από τώρα μέχρι το 2020 και θα πρέπει επίσης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τα υπόλοιπα στοιχεία ε, για να απαντήσουμε στις μεταναστευτικές πιέσεις ε, στον τομέα του ασύλου και της ε, ένταξης και των κονδυλίων ασφαλείας και τις δαπάνες που σχετίζονται με τα αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Επομένως, υπάρχουν δύο στιγμές στον προϋπολογισμό θα έλεγα. Στην αρχή θέλουμε μια εκτίμηση πιο επακριβή για τις προβλέψεις για την επόμενη χρονιά, κάτι το οποίο θα γίνει για τον προϋπολογισμό του 2017 και από εκεί και πέρα ε, για το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020 θα πρέπει να γίνει μια προβολή μέχρι και το 2020 και κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση των ε, ε, των πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε και τα διαθέσιμα κονδύλια στις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά αργότερα για το 2017 ίσως ε, θα μπορέσουμε να το έχουμε αυτό στο σχέδιο προπολογισμού και στις προβλέψεις που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τομά είπε ότι ανησυχεί λίγο για την αβεβαιότητα που εξέφρασα κι εγώ. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε λίγο από πού προκύπτει αυτή η αβεβαιότητα. Το παράδειγμα σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου. Αυτή τη στιγμή Παρακολουθούμε βέβαια και πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις επόμενες ομάδες, ε, εβδομάδες. Έχουμε δύο στόχους για την ε, μεταρρύθμιση και ο ένας από αυτούς δεν είναι πραγματικός στόχος. Ο πρώτος στόχος είναι να παραμείνει η κατάσταση ε, ευρύτατα ως έχει, να έχουμε δηλαδή τα βασικά κριτήρια, τα οποία σημαίνει ότι η Ελλάδα, εάν συνεχίσουν οι αφήξεις όπως έχουν αυτή τη στιγμή, θα βρεθεί ενώπιον μιας αφόρητης κατάστασης. Μετά, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δεύτερο κριτήριο στο κανονισμό του Δουβλίνου, αλλά εκεί θα αναγνωρίζουμε ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τέτοια ότι, ώστε χρειάζεται ένα σύστημα ε, με κρίσης, διότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τις παρούσες ε, ροές. Αυτή θα σημαίνει ότι θα υπάρχει ήδη ένα σύστημα μετεγκατάστασης ε, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, υπάρχει δηλαδή αυτό το οποίο είναι διαθέσιμο τουλάχιστον για το προσεχές μέλλον. Και από εκεί και πέρα η επόμενη επιλογή θα ήταν να ξεκινήσει πολιτική μια κατάσταση όπου θα υπάρχει μια μόνιμη κλίδα κατανομής ε, που θα συζητηθεί στο Δουβλίνο και οικονομικά φυσικά θα είμαστε σε τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Αυτό σας το δίνω ως παράδειγμα για να σας εξηγήσω αυτό που είπα λίγο αφαιρημένα στην παρέμβασή μου. Πρέπει να περιμένουμε λίγο τις επόμενες εβδομάδες να δούμε πώς θα διαμορφωθούν και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό φυσικά θα έχει συνέπειες και για τους υπολογισμού που θα κάνουμε εμείς στον προπολογισμό. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να σας δώσω αυτό το παράδειγμα και φυσικά θα μπορούσαν να υπάρξουν και πολλά άλλα. Ευχαριστώ. Ωραία. και για την ε, κατανομή αυτών των χιλίων ε, ε, συνοριοφυλάκων, ποιοι θα είναι στη Βαρσοβία, ποιοι θα είναι στα σύνορα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει βέβαια να κατανοήσετε ότι αυτή είναι ακόμα η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Το σχέδιο είναι οι περισσότεροι από αυτού να εργάζονται στην έδρα μα. Συνεχώ όμω, στι επιχειρήσει μα και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και σε κάποιε άλλε περιπτώσει έχουμε μέλη του προσωπικού μα που ε, ε, πηγαίνουν εκ περιτροπή για το συντονισμό των εργασιών και αυτό θα αυξηθεί. Ε, χονδρικά να σας πω ότι από αυτούς τους ε, χιλίους ή εξακοσίους επιπλέον ε, νέους υπαλλήλους θα έχουμε περίπου 100 με 200 αυτής της μορφής, οι οποίοι εκ περιτροπής θα εργάζονται επιτόπου τόπου στα σύνορα για να γίνεται συντονισμός των διαφόρων καθηκόντων και να υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των σύνορων. Αυτές είναι οι χονδρικές εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή, διότι ακόμα είμαστε στο ε, στάδιο του προγραμματισμού και θα δούμε ανάλογα με το αποτέλεσμα του νέου κανονισμού και των νέων καθηκόντων του οργανισμού. Ευχαριστώ. Ο Μαρζή. Α, ο Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και χαιρετίζω τις προσπάθειες της Κομισιόν για την παρουσίαση που έγινε. Ε, υπάρχουν πέντε στόχοι εδώ που καταδεικνύουν την αποτυχία των πολιτικά ηθινόντων της Ευρώπης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Φαίνεται ότι επενδύεται πολλές ε, ελπίδες στο συμβούλιο το οποίο ξεκινάει σήμερα με ένα δείπνο, αλλά εάν ε, ε, αλλά από ό,τι φαίνεται απλώς θα διπνήσουν και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απόφαση σήμερα και θα πρέπει να περιμένουμε το μήνα Μάρτιο ενώ πραγματικά η κρίση υπάρχει σοβή και πραγματικά υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα πέντε αυτά σημεία, ακούω τα όσα λέτε όσον αφορά τη βοήθεια προς την Ιταλία και την Ελλάδα. Αλλά όσον αφορά τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, θα πρέπει επίσης για να είμαστε αντικειμενικοί να υπογραμμίσουμε την έλλειψη της υποστήριξης εκ μέρους του προπολογισμού ε, όσον αφορά τη βοήθεια προς την Ελλάδα και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε επίσης την έλλειψη αλληλεγγύης έναντι αυτών των χωρών ε, γιατί υπάρχει αυτό το παράλογο ε, ε, που φτάνει μέχρι τον παραλογισμό να λέμε ότι θα πρέπει να βγει η Ελλάδα από τη ζώνη Σέγγεν. Και πραγματικά εδώ διατυπώνω έναν προβληματισμό. Τον περασμένο αιώνα η ελευθερία ήταν πραγματικά να πέσουν τα τείχη. Και βλέπουμε με την κρίση αυτή ότι σήμερα ε, με την προσπάθεια να εψωθούν νέα τύχη δηλαδή να τεθεί ένα αμφιβόλο το Σέγγεν ε, προσπαθούμε να διανοηθούμε τη μελλοντική πρόοδο και εξέλιξη. Και όσον αφορά τον τελευταίο στόχο, είναι απολύτως προφανές ότι πρόκειται για ένα στόχο τον οποίο συμμεριζόμαστε, αλλά ο οποίος ε, συνεπάγεται μια εις βάθος ε, αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής πολιτικής αν θέλουμε να αλλάξουμε τους όρους αντιμετώπισης των χωρών της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Ευχαριστούμε, δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, άρα θα επωφεληθώ για να, θέσω προσωπικά, για να αναπτύξω προσωπικά μερικές ε, σκέψεις. Και πάλι ε, αυτό το οποίο επιτελεί η Κομισιόν και η Frontex είναι πραγματικά αξιοσημείωτα. Αλλά στις στατιστικές τις οποίες αναφέρατε, παρόλα αυτά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια δυσαναλογία μεταξύ των στόχων που εκφράζονται και στόχων και της πραγματικότητας από την άλλη. Γιατί κάθε μέρα ε, φτάνουν ε, από 3 5 ε, πρόσφυγες και από το Σεπτέμβριο έχουν επιστραφεί 650 άτομα. Βεβαίως αυτό είναι θετικό γιατί επιτρέπει ε, στις κυβερνήσεις ε, να κάνουν δηλώσεις αλλά δεν ρυθμίζεται κανένα απολύτως πρόβλημα. Επίσης η μετακατάσταση και το σχετικό πρόγραμμα είναι απόλυτη αποτυχία. Και κάθε χώρα μέλον έχει, ε, μέλος έχει τη δική της ε, ερμηνεία όσον αφορά τη χορήγηση ασύλου σε ορισμένες χώρες. Μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν άμεσα, αλλού μετά από ένα χρόνο, τα επίπεδα αποδοχών διαφέρουν, οι συνθήκες υποδοχής διαφέρουν και οι πρόσφυγες ε, κάνουν τη δική τους επιλογή και έχω κατά νου αυτά τα οποία προσπάθησε η πρόεδρος του Λουξεμβούργου ε, προβάλλοντας ε, προς την κοινή γνώμη το θέαμα της άφηξης ενός ε, αεροπλάνου γεμάτου από σύρους, οι οποίοι όμως δεν πήγαιναν στο Λουξεμβούργο και υπήρχαν όλες οι εκπρόσωποι όλων θεσμικών οργάνων, πολύ θεαματικό εγχείρημα αλλά που δείχνουν ότι δεν είναι καθόλου προφανές το εγχείρημα της μετεγκατάστασης και τελικά περιορίζεται σε ελάχιστους. Όσον αφορά τη Frontex, αυτό το οποίο με καταπλήσει είναι ότι πραγματικά βάζουμε πολύ λίγα χρήματα στα σύνορα και τα περισσότερα επενδύονται στην ένδρα, σαν να πρόκειται για την προσπάθεια οικοδόμησης μιας κεντρικής έδρας, παρόλο που είναι παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να προσελκυστούν ε, συνεργάτες. Ε, ε, ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Frontex έχει την έδρα στη Βαρσοβία η οποία ακόμα δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία. Δηλαδή, τι είναι το θέμα της έδρας, είναι το ζήτημα του φορολογικού καθεστώτος, της εκπαίδευσης των παιδιών, τι γίνεται με το θέμα αυτό της έδρας. Ε, και επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι έχουμε ανάγκη μια αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τον αντίκτυπο στο μέλλον. Ε, το σπίτι μας καίγεται, αλλά θα περιμένουμε πολλά χρόνια για να φτάσουμε στους χίλιους εργαζόμενους. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά είναι σουρεαλιστικά και διερωτάται κανείς ε, ποια είναι, ε, πώς κυβερνιέται αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της νομικής βάσης θα μου απαντήσετε, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε γραφειοκρατικές και τεχνοκρατικές στάσεις, τάσεις που περιπλέκουν τα μέγιστα το, ε, την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Ε, βεβαίως πώς μπορεί να είναι κανείς αποτελεσματικός στο πλαίσιο τέτοιων ε, καταναγκασμών, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Ωραία λοιπόν, εάν θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας, δεν ξέρω, στρέφουμε στους συναδέλφους, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, η ψηφορία προβλέπεται το μεσημέρι, και στις 11.40 ε, έχουμε μια ε, ανακοίνωση. Άρα θα κλείσει, η, θα ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή στις παρα 25. Βεβαίως, αν θέλετε κάποιες ευκρινήσεις και ερωτήσεις, έχουμε το χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, για να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μια ε, υπηρεσία ακτοφυλιακή και συνοριοφυλιακή. Ε, Σαφώ και υπάρχει και δημόσιο νομικό σχεδιασμό που σχετίζεται με την πρόταση και που έχει σταλεί στην αρμόδια αρχή, στι νομοθετικέ αρχέ και στο Κοινοβούλιο δηλαδή και η συγκεκριμένη εκτίμηση του κόστους και του καταμερισμού του κόστους είναι στο δημοσιονομικό δελτίο το οποίο προβλέπει και το ε, διάστημα μέχρι το 2020. Δεν το έχουμε συμπεριλάβει στις διαφάνειές μας γιατί είναι αρκετά αναλυτικό, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να σας ξαναστείλουμε το δελτίο ε, για να μην έχετε την εντύπωση ότι θέλουμε να σας ε, κρύψουμε πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. Όσον αφορά το θέμα της εφαρμογής ε, της ε, μείωσης ε, του 5% στο προσωπικό του Frontex. Ξέρετε ότι υπάρχει απόφαση η οποία περιλαμβάνεται στη διοργανική συμφωνία που προβλέπει ότι πρέπει να μειωθεί κατά 5% το προσωπικό και οι θέσεις οι οποίες ε, δίνονται και στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς και στις υπηρεσίες. Επομένως ξεκινά ε, μια διαδικασία που είναι θέμα προϋπολογισμού και έχει ε, συσταθεί και μια διοργανική ομάδα. Οι αποφάσεις για τον καταμερισμό των θέσεων γίνονται σε μια αιτήσια διαδικασία κατόπιν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την έγκριση φυσικά των δημοσιονομικών αρχών. Για την περίπτωση του Frontex έχουμε μία αύξηση των υπαλλήλων που θα προκύψει. Επομένως νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να δούμε και το συνολικό αποτέλεσμα που θα έχουμε στο τέλος, γιατί θα υπάρχει μία ουσιαστική αύξηση εκεί. Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο στο Ματίας. Ευχαριστώ. Να απαντήσω με τη σειρά που ετέθησαν τα ερωτήματα. Μιλήσατε για την έλλειψη των ε, χρηματοπιστωτικών ε, πόρων. Είναι καλό να ε, καταγραφεί αυτό όντως. Να σας θυμίσω την οικονομική στήριξη που έχει δώσει η Ευρώπη στην Ελλάδα μέχρι τώρα. Η Ελλάδα στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων για το άσυλο και την ολοκλήρωση και στα πλαίσια του Ταμείου για την ασφάλεια φτάνουν τα 5,9 εκατομμύρια για την ε, περίοδο 2014-2020. Τα, τα, κονδύλια που αποδόθηκαν στην Ελλάδα για την ενίσχυση της προσπάθειας να ενισχύσει τις αποδομές της όπως ε, οι υποδοχές, ε, λήψη αποφάσεων, ολοκλήρωση, επιστροφές, συνοριακή έλεγχη, εποπτεία, αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας και των λαθρεμπόρων και ασφάλεια. Ε, ε, έχει ως εξής. 33 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015. Επίσης, άλλη μια πληρωμή θα γίνει σύντομα με 36 εκατομμύρια ευρώ ως προχρηματοδότηση για το 2016. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει ουσιαστική πήγουσα στήριξη περίπου 145 εκατομμυρίων ευρώ στα πλαίσια του ΑΜΙΦ και του ISF για την Ελλάδα είτε ε, άμεσα στις ε, ε, ελληνικές αρχές, είτε μέσω διεθνών οργανισμών για εφαρμογή δράσεων στις, στη χώρα αυτή το τελευταίο έτος. Στην Ελλάδα, ας πούμε, πρόσφατα μια, είχαμε μια συμφωνία με την υπατερμοστία του ΟΗΕ για 80 εκατομμύρια, για 80 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής στην Ελλάδα. 6,3 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί επίσης για ε, στήριξη επίγουσα και αν δούμε και την ε, στήριξη που υπάρχει στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας και την ε, επίγουσα στήριξη που έχει δοθεί στην Ελλάδα μέχρι τώρα, η Ελλάδα είναι ο πρώτος δικαιούχος ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Home με περίπου 255 εκατομμύρια ευρώ. Να πω επίσης ότι σε σχέση με την, ενίσχυση, με την με κατασκευή των hot spots και η ΆΖΟ και η Frontex ε, είναι επιτόπου στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται και εμεί ω Γενική Διεύθυνση Home έχουμε τέσσερι συναδέλφου στην Ελλάδα και τέσσερι συναδέλφου στη Ρώμη για να εφαρμόσουμε τα προγράμματα επανεγκατάσταση και βεβαίως θα συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη στην Ελλάδα που βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να πω όμως ότι η Ελλάδα τώρα πρέπει να αρχίσει να χρησιμοποιεί τους πόρους που είναι διαθέσιμοι και να εφαρμόσει τα εθνικά της προγράμματα. Τελευταίο σημείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει και τα διαρθωτικά ε, ταμεία για την δημιουργία ε, δυνατοτήτων υποδοχής στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για μέτρα που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη. Και ε, από εκεί υπάρχουν κονδύλια λοιπόν. Αυτά γενικώ για να σας ε, δείξω τι σημαίνει αλληλεγγύη και πώς την ε, δίνουμε προς την Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, εσείς θέσατε κάποια ερωτήματα για την μετεγκατάσταση. Ε, Βεβαίως ε, είπα ότι το, η εφαρμογή δεν είναι ε, ε, επικοδομητική, έτσι το βλέπει η Κομισιόν. Να πω όμως το εξής, να μην το ξεχάσουμε κιόλα. τα προγράμματα αυτά διαρκούν δύο χρόνια. Ο λόγος είναι ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ πιο σύντομη. Αλλά μετά υπήρξαν αρκετά κρατημέλη που είπαν και δικαίως ότι πρέπει να κατασκευάσουν αυτά τα κέντρα, τις υποδομές. Υπάρχουν κάποια κράτη που για να κάνουν τη μετεγκατάσταση δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουν ε, ε, κέντρα υποδοχής ε, μεταναστών ή προσφύγων. Γι' αυτό ο συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε στο τέλος ήταν ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να ισχύει για δύο χρόνια. Οπότε Εντάξει, τα κράτη-μέλη λένε ότι δεν έχουμε μεταγκαταστήσει κανέναν πρόσφυγα μέχρι τώρα, αλλά θα το κάνουμε στο μέλλον. Και επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να σας πω ειλικρινώς, είναι ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, αλλά σε πολλές φορές ε, ε, χρειάζεται συμφωνία και με τους πρόσφυγες. Ένα τρίτο πρόβλημα που πρέπει να σας αναφέρω είναι ότι ε, αυτά τα προγράμματα ανακατανομής τα προτείνουμε για να δημιουργήσουμε διασπορά σε κάποια και αυτό οδηγεί ακριβώς και στην, ε, στο δισταγμό που δείχνουν οι πρόσφυγες να πάνε σε χώρες που δεν ξέρουν. Δεν θέλει κανείς να είναι ο πρώτος ε, που θα πάει στην Εστονία. Είναι προτιμότερο να πάει εκεί που είναι και οι άλλοι 5.000, στη Γερμανία για παράδειγμα. Ε, οπότε μόλις ξεκινήσουν να γίνονται οι πρώτες ανακατανομές τότε θα υπάρξει έτσι ε, πιο μεγάλη θέληση και από τους ίδιους τους πρόσφυγες αλλά προφανώς η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιητική. Όπως είπα, το πρόγραμμα αυτό της επανεγκατάστασης ε, λειτουργεί σχετικά καλά όπως είπα. Μιλήσατε για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Να θυμίσω λίγο την νομική κατάσταση. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να, έχει, να επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας μετά από 9 μήνες. Έτσι έχει το νομικό πλαίσιο. Τα κράτη-μέλη βεβαίω ε, αυτό μπορούν να το κάνουν και πιο νωρί αν ε, το επιθυμούν. Επίσης αναφέρατε, και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο, ότι οι μετανάστες ε, διαλέγουν τελευταίο στις χώρες που θα πάνε. Σωστή είναι αυτή η αξιολόγηση. Ο λόγος είναι ότι προς το παρόν δεν έχουμε ένα καλά λειτουργών σύστημα Δουβλίνου. Δεν δουλεύει δίκαια πλέον το Δουβλίνο και γι' αυτό θα πρέπει σύντομα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για ένα νέο σύστημα Δουβλίνου. Και το πιο σημαντικό ακόμη, όπως είπα ήδη, είναι ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τους νομικούς κανόνες με συνέπεια, γιατί αλλιώς δεν θα λειτουργήσουν. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο τώρα στο συνάδελφο από τη Frontex. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω για τα θέματα επιστροφών, για τις προκλήσεις που υπάρχουν, κάποια σημεία για, την, για το προσωπικό και για τα κεντρικά και για τα αρχηγεία. Οι προκλήσεις για τις ε, επιστροφές λαθρομεταναστών ή παραμένως διαμενόντων ε, τρεις είναι οι βασικές προκλήσεις. Καταρχάς, έχουμε πολλά άτομα στα σύνορα που πρέπει να ταυτοποιηθούν. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση η πρώτη. Συνήθως τα άτομα αυτά, όπω είπατε 2.000 τη μέρα καμιά φορά και ίσως και περισσότεροι, δεν έχουν χαρτιά. Δεν έχουν ταυτότητες, Οι περισσότεροι λένε ότι είναι από τη Συρία. Έχουμε το προσωπικό μας εκεί και τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που ξέρουν τη γλώσσα, πολιτιστικούς ε, ε, συμβούλους τους ονομάζουμε, για να μιλήσουν με τους ανθρώπους αυτούς στη μητρική τους γλώσσα, για να μπορέσουν να καταλάβουν αν όντως τα άτομα αυτά είναι από την Ανατολική Συρία, από την Νότιο Συρία, από την Παλαιστίνη, από το Πακιστάν. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση. Πώς ταυτοποιούμε αυτά τα άτομα. Αν καταφέρουμε να τα ταυτοποιήσουμε μαζί με τις ελληνικές αρχές, μετά καταγράφονται. Δεύτερη, ε, δεύτερη πρόκληση. Μετά αυτή την καταγραφή, την καταχώρηση, πηγαίνουν σε δύο διαφορετικές διαδικασίες. Μία είναι η επιστροφή για αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα να μείνουν, δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Και η άλλη ομάδα είναι αυτή που μπαίνουν στην διαδικασία παροχής ασύλου, όπου υπάρχει όντως ανάγκη παροχής διεθνούς προστασίας. Αυτή η διαδικασία παίρνει το χρόνο της. Και μετά αυτό φεύγει από τα χέρια της Frontex. Είναι θέμα του κράτους μέλους και της ΕΑΖΟ να το τρέξουν, να το διεκπαιρεώσουν. Μετά έχουμε τον, ένα χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο αυτά τα άτομα κάπου πρέπει να μπουν, πρέπει να στεγαστούν κάπου. Πρέπει να τους δοθεί ιατρική περίθαλψη αν χρειάζεται. Πρέπει να τους δοθεί ε, κατάλημα. Πρέπει να τους δοθεί τροφή. Αυτή είναι η Επόμενη πρόκληση. Δεν έχουμε επαρκείς ε, εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, στα νησιά αυτά. Οπότε, δεύτερη πρόκληση. Μετά από δύο εβδομάδες εξαφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε πού είναι ο κύριος Τάδε ή ο κύριος Δίνα. Έχουν εξαφανιστεί. Αυτή είναι ακόμα μια μεγάλη πρόκληση. Ε, ταυτοποίηση και ε, στέγαση και μετά τελικά. Αν όντω έχουμε ένα άτομο που πρέπει να επιστρέψει, πρέπει να έχουμε μια χώρα η οποία θα πρέπει να, τον, να, θέλει να τον παραλάβει. Και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Πού επιστρέφουν οι άνθρωποι. Αν η χώρα προέλευσης δεν θέλει να τους ε, υποδεχθεί, αν η χώρα προέλευσης δεν θέλει να του δώσει ε, ταξιδιωτικό έγγραφο, γιατί χρειάζεται κάποιο είδος ταξιδιωτικό έγγραφο για να επιστρέψει κάποιος, τότε το πρόβλημα ε, μεγαλώνει. Γι' αυτό είπαμε ότι εμεί πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο. Αλλά αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος, γιατί η τρίτη αυτή χώρα θα πρέπει να συμφωνήσει να δεχτεί αυτά τα ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά ε, ε, έγγραφα για λόγους, ε, για σκοπούς επιστροφή. Υπάρχουν λοιπόν και στα πλαίσια τη επιστροφή πολλέ προκλήσει. Λέμε ναι, πρέπει να επιστρέψουν πάνω από 600 το χρόνο, περισσότεροι, αλλά όπω σα εξηγώ, δεν είναι στην πράξη τόσο απλό να γίνει αυτό. Τώρα, να περάσω στο δεύτερο ερώτημα. Ίσως ε, να μην ήταν απόλυτα σαφές αυτό που είπα. Τα, ο προσωπικό της Frontex δεν κάνει τη δουλειά αυτή στο, στα, στα σύνορα. Έχουμε και το καθήκον να έχουμε και τους συνοριοφύλακες που θα πρέπει να τους εκπαιδεύουμε, που θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να έχουν και τη θέληση να δουλέψουν σε αυτές τις ε, συντονισμένες επιχειρήσεις. Έχουμε 3.000 συνοριοφύλακες. Συνοριοφύλακες που δουλεύουν καθημερινά στα κράτη τους και μετά από κάποια περίοδο προειδοποίησης που τους δίνουμε εντάσσονται στις ε, μικτές επιχειρήσεις τις οποίες ε, διεξάγει η Frontex. Έχουμε λοιπόν κάποιους, κάποιες χιλιάδες συνοριοφύλακες. Αυτοί είναι αυτοί που κάνουν ε, τη δουλειά. Το δικό μας το προσωπικό ουσιαστικά το συντονισμό αναλαμβάνει, το συντονισμό της δουλειάς. Έτσι δουλεύει η Frontex. Εμείς έχουμε έτσι μια βάση δεδομένων ας πούμε, ονομάτων συνοριοφυλάκων που μπορούν να κάνουν τη δουλειά αυτή και όταν τους χρειαζόμαστε τους καλούμε, χρηματοδοτούμε τις ε, επιχειρήσεις και τους βάζουμε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει στα νησιά αυτά στην Ελλάδα. Γι' αυτό τα δικό μας το προσωπικό δεν ε, είναι είτε τόσο πολύ είτε τόσο συχνά επιτόπου. Για τις συμφωνίες ε, για τα αρχηγεία. Ξέρετε ότι για να διαπραγματευτεί κανείς πρέπει να έχει και έναν συνομιλητή. Έχουμε θέσει τρία ερωτήματα στις πολωνικές αρχές για να ξεκινήσουμε να διαπραγματευόμαστε. Εστήριξη για τη στέγαση καταρχάς. Θα θυμάστε ότι η Frontex καταβάλει 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να ενοικιάζει τις εγκαταστάσεις στη Βαρσοβία. Δεύτερον, θέλουμε να έχουμε κάποιο εχέγγυο ότι το προσωπικό, τα παιδιά του προσωπικού θα έχουν ε, ε, εκπαίδευση πολυγλωσσική, ευρωπαϊκής ε, νοοτροπίας. Και επίσης θέλουμε να υπάρχει σαφήνεια για το καθεστώς μας. Εμείς τι, τι θεωρούμαστε. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Αυτά είναι τα τρία ερωτήματα που έχουμε θέσει και σε αυτά έχουμε κολλήσει, πρέπει να πω. Δεν έχουμε πολύ πρόοδο. Αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος ε, διατάζει, ποιος ε, κάνει κουμάντο. Ε, δίνουμε κονδύλια στην Πολωνία κάθε χρόνο. Η Πολωνία έχει κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν τηρεί. Είναι εκπληκτικά όλα αυτά τα πράγματα. πώς θα τα εξηγήσουμε εμείς αυτά στους πολίτες μας όταν μας ρωτήσουν τι γίνεται. Πραγματικά με σοκάρουν αυτά. Δεν πάντων, μην εκνευρίζομαι. Δύο ε, άτομα έχουν ζητήσει το λόγο, σύντομα, γιατί φτάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Ο κύριο Ρούμπικ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά θα με ενδιαφέρει να μου πείτε πώς διαμορφώνεται η συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Frontex και πώς συντονίζεται. Και ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Deuxième intervenant, Madame η κυρία ε, Λυπούμε, αλλά μερικές φορές ε, αργεί μετάφραση. Κατάλαβα καλά ότι η Ελλάδα έχει, ε, θα πάρει 66 εκατομμύρια από το Ταμείο για το προσφυγικό. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δουλειά σας, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε μέσω μιας έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου έχουμε την πληροφορία ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πάνε καλά, δεν λειτουργούν. Ε, τι, τι ελπίδες έχουμε ότι θα λειτουργήσουν και ότι τα πράγματα θα φτάσουν εκεί που πρέπει να πάνε. Και εκ μέρους της Frontex ε, ποιος το ελέγχει αυτό και πώς, με ποιο τρόπο. Οι ερωτήσεις ήταν σύντομες, ε, άρα πρέπει και εσείς να είστε σύντομοι στις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το Frontex και το ΝΑΤΟ, μια πολύ σύντομη απάντηση. Δεν υπάρχει ακόμα τέτοια συνεργασία. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ε, δημιουργήσουμε τη συνεργασία αυτή. Στη συνέχεια θα γνωρίζουμε περισσότερα. Ο κύριος Ζωέλ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση της κυρίας Κρέσλε 655. 650 εκατομμύρια ευρώ συνολικά ε, καταμορισμός των εθνικών προγραμμάτων και κατεπίγουσα βοήθεια έχουν καταβληθεί. Όπως ε, σας είπα στην παρουσίασή μου, πέραν ε, ενός ε, τα hot spot ε, στην Ελλάδα είναι πλέον σε λειτουργία. Επιτέπου υποστηρίζουμε τους Έλληνες για την εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει για να υπάρχει ένα συνολικός ε, συντονισμός ε, η Επιτροπή και το SRSS. Ε, και να σας πω το εξής. Αν σκεφτείτε τι ροές είχαμε στην Ελλάδα, περίπου 850.000 άνθρωποι έφτασαν στην Ελλάδα πολλοί από αυτούς εξαφανίστηκαν. Και αν το ε, συνυπολογίσετε αυτό με βάση τον πληθυσμό της Γερμανίας, θα πρέπει να το πολλαπλασιάσετε επί 8 και θα δείτε ότι έχουμε πάνω από 6 εκατομμύρια ε, πρόσφυγες. Ε, ε, αυτή είναι η κλίμακα ε, των μεταναστών που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να υπάρξει και υποστήριξη. Και όσον αφορά την, τον έλεγχο. Είναι μια πολύ συνηθισμένη διαδικασία. Θα γίνονται έλεγχοι και από το ελεκτικό συνέδριο. Υπάρχει μια νέα δομή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε αρχίσει να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμα, λοιπόν, για να συνοψίσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτο συμπέρασμα, ακόμα βέβαια πολύ δειλά, Νομίζω ότι εκπροσωπώ όλα τα μέλη τη Επιτροπής προπολογισμών, όταν λέω ότι για τον τίτλο 4 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένο για τις εξηγήσεις που δόθηκαν για τις ε, ε, ε, εξωτερικές δράσεις παρά το γεγονός ότι η κυρία Καλβίνιο μας είπε και μας έδωσε πολλά στοιχεία νομίζω ότι μπορώ να πω ότι τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι εξοργισμένα διότι όλα τα επιχειρήματα τα οποία παρουσιάστηκαν για να αιτιολογηθούν κάποια εξωτερικά ε, μέσα ε, στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά το συντονισμό και την ευελιξία θα μπορούσαν κάλλιστα να συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και στην διάμεση αναθεώρηση. Πόσο μάλλον που αυτά τα μέσα και αυτή η ανάλυση δεν αντιμετωπίζουν τελικά την κατεπίγουσα κατάσταση για την οποία υποτίθεται ότι χρησιμοποιείται ο ίδιος ο προπολογισμό της Ένωσης. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η προστιθέμενη αξία τους λοιπόν, διότι δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τα χρήματα δεν φτάνουν απαραίτητα εκεί που θα έπρεπε να φτάσουν, όπως είπε και ο Πρόεδρος και τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας που ε, ήταν στην ε, αποστολή στην Τουρκία. Και επιπλέον, τα ίδια χρήματα, τα ίδια ποσά τα οποία δαπανώνται σε αυτά τα εξωτερικά κονδύλια που θα ε, ε, μπορούσαν να δαπανηθούν αν ήταν στον προπολογισμό της Ένωσης, μπορεί και περισσότερα, διότι το κόστος διαχείρισης, όπως είπα και προηγουμένως, αυξίζουν ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι αυτά γίνονται εκτός. Ε, η Επιτροπή μας λοιπόν είναι εξοργισμένη και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να εξαγριωθούμε και να επαναστατήσουμε για αυτά τα οποία μας είπατε, διότι θεωρούμε ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα, δεν υπάρχει κατάλληλη προβολή, δεν υπάρχει διαφάνεια και δεν υπάρχει κοινοβουλευτικό έλεγχο εν τέλει. Όσον αφορά τον τίτλο 3, εδώ η ανησυχία από πλευρά μου και νομίζω ότι το ίδιο άκουσα και από τις παρεμβάσεις ε, των συναδέλφων είναι πολύ μεγάλη φαίνεται ότι δεν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες αξιολογήσεις των αναγκών του 2017. Εντάξει, αυτό κατανοητό και το είπα και στις ερωτήσεις μου προηγουμένως, αλλά ε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα, τα οποία είναι πολύ ανεσυχητικά. και το πιο σοβαρό δεν είναι αυτά που ακούσαμε, αλλά ότι μας δίνεται εντύπωση ότι τα μέσα τα οποία έχουν προβλεφθεί ή μας ανακοινώθηκαν δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή από τις πέντε αποστολές που μας υπενθυμίσατε, κύριο Ελ, και που ε, με τις οποίες συμφωνούμε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, ε, δεν φαίνεται να υπάρχουν τα κατάλληλα κονδύλια για να ε, υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν. Και επίσης δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι τα κονδύλια είναι κατάλληλα, αλλά οι ανακοινώσει του Συμβουλίου φαίνεται να είναι τελείως διαφορετικές από τα αρχικά ποσά τα οποία υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιηθούν. Όταν μας λένε με ε, μεγάλα λόγια ότι θα έχουμε συνοριοφύλακες, κανείς δεν σκέφτεται ότι θα έχουμε 100 συνοριοφύλακες που θα ε, εργάζονται επιτόπου σε όλα τα σύνορα της Ένωσης. Ε, σκεφτόμαστε πολύ πιο σημαντικές δυνάμεις. Και μετά, για την Ελλάδα θεωρώ ότι η συζήτηση είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη. Ε, ο τρόπος με τον οποίο μας τα παρουσιάζεται μου δημιουργεί προβλήματα. Αλλά μου υπόψη ότι υπάρχει ακόμα η Σέγγεν και ότι κατά συνέπεια πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας ε, ε, γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε κατά την άποψή μου να λέμε ότι α, δίνουμε βοήθεια στην Ελλάδα. Δεν δίνουμε βοήθεια στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να στήσουμε ευρωπαϊκά σύνορα. Έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Καμία χώρα δεν είναι υπεύθυνη για τα γεωγραφικά της σύνορα και η Ελλάδα δεν είναι υπεύθυνη για το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη πόρτα εισόδου ε, το, από τη Μέση Ανατολή και δυστυχώς ε, από τους πρόσφυγες του πολέμου της Συρίας. Και πολλό δε μάλλον το ίδιο ισχύει και για την Ιταλία. Ε, δεν φταίει η Ιταλία που είναι μια χερσόνησος που επιτρέπει την πολύ εύκολη πρόσβαση από τις αφρικανικές ακτές από και δεν είναι το ίδιο με την Πολωνία παραδείγματος χάλη Πιστεύω ότι χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση για τα ευρωπαϊκά σύνορα και να μην υπάρχει απλώς ενίσχυση. Ε, αυτή τη στιγμή δυστυχώς αυτό που έχουμε δεν είναι ευρωπαϊκή διάταξη. Ε, το ακούσαμε και από το Διευθυντή του Frontex. Ε, πρόκειται για μια διάταξη η οποία προσπαθεί να συντονίσει αυτά τα οποία υπάρχουν και τίποτα περισσότερο. Και νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι μεταξύ των ανακοινώσεων και των πραγματικών μέσων που δίνονται για την επιχειρησιακή εφαρμογή αυτών των αποστολών που ανακοινώθηκαν, υπάρχει ένα χάσμα, το οποίο χάσμα με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κλείσουμε. Ευχαριστώ κυρία τομά, Ευχαριστώ τους ε, προσκεκλισμένους, τον κύριο Πρέζα, τον κύριο Ελά, τον κύριο Βένσολα, την κυρία Καλβινιό η οποία έφυγε. Καταλάβατε ότι υπάρχει μια κάποια διαμαρτυρία από πλευράς μας. Ε, το κάποια είναι φημισμός. Ε, θα θέλαμε η κυρία Γεωργίευα να μπαίνει στον κόπο να μας ενημερώνει επισήμως και όχι με μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση για ουσιώδη θέματα. Ε, είναι και ένδειξη ε, καλή συμπεριφορά ε, μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα τέλο εποχή όσον αφορά τον προπολογισμό. Έχουμε αρχίσει και φτάνουμε και στα πλαίσια του γελίου ορισμένε φορέ διαπιστώνω ότι σταμάτησαν προς στιγμή οι εργασίες. Έπρεπε να έρχει ο κύριος ε, Μότι για να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα των ιδίων πόρων, αλλά επειδή ε, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το θέμα του Βρετανικού Δημοψηφίσματος, ε, το έχουμε καθυστερήσει αυτό. Το θέμα είναι θα μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε αν δεν ε, ολοκληρωθεί το θέμα του Δημοψηφίσματος. Αν μπορούσαμε να επιταχύνουμε λίγο με το Βρετανικό ζήτημα, ίσως θα μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριοι και κυρίες και καλό κουράγιο. Ξέρουμε ότι σας περιμένει δύσκολη δουλειά και ότι κάνετε ό,τι μπορείτε. Αλλά έχουμε δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε και το κάνουμε. Και τώρα, έκθεση της κυρίας Χέλγα Τρούπελ, η οποία έχει κάνει συντάξει μια γνωμοδότηση για τον έλεγχο του Μητρώου και τη σύνθεση των ε, Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων. Ε, τώρα θα μιλήσουμε για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και θα ασχοληθεί με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή έχει πάνω από 100 ομάδες εμπειρογνωμόνων που παρέχουν τις συμβουλές της στην διαδικασία νομοθέτησης. Και έχουμε, ασκούμε εδώ την κριτική ότι υπάρχει μια διαφάνεια σε αυτές τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και η σύνθεσή τους δεν είναι αρκετά ισορροπημένη. Γι' αυτό ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμών αποφάσισε ήδη το 2011 και το 2014 να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα εν σχέση με το τι επιθυμούμε. Και τώρα έχουμε μια πρόσφατη μελέτη ε, που ανατέθηκε από την Επιτροπή Προπολογισμών που διαπιστώνει ότι υπάρχει διαφάνεια και έλλειψη ισορροπίας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε ως, ε, αυτό το οποίο θέλαμε ως μεταρρύθμιση μέχρι στιγμής δεν έχει ε, επιτευχθεί και η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια υπογραμμίζει στις συστάσεις της να αυξηθεί η διαφάνεια στις επιτροπές, στις ομάδες Και τώρα συνειδητοποιούμε ότι η Επιτροπή εξαγγέλει ότι θα προχωρήσει μεταρρυθμίσεις, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι εν σχέση με τις ε, προϋποθέσεις που θέτουμε. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να τηρούνται οι οριζόντιοι κανόνες γιατί στη μελέτη κατέστη σαφές ότι έχουμε μία αύξηση ε, μια μείωση των μη ε, οικονομικών ε, μελών. θέλουμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αναλάβει δράση όταν έχουμε να κάνουμε με ομάδες που εκπροσωπούνται και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη θέση τους όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη ή ε, το να προστρέξουν σε ορισμένα άτομα που γνωρίζουν άμεσα περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό θέλουμε η συνεργασία με τις ομάδες αυτές ε, να μπορεί να επιτελείται. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τι θα κάνει η Επιτροπή και κατά πόσο θα ικανοποιήσει τους όρους μας και λέμε ότι αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι μας θα πάμε στα αποθεματικά ε, ούτως ώστε να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις για το 2017. Ε, αυτή είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση. Η κυρία Γκρέσλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω απλώς ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό πρόβλημα με την έκθεση πρωτοβουλίας γιατί η Επιτροπή εντωμεταξύ μας ε, είπε ότι προσεχώς θα υπάρξουν νέες οδηγίες για το ζήτημα της σύνθεσης των, των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Ο εισηγητής γι' αυτό θέλει να συνομιλήσει με την Επιτροπή για να κατά πόσο θα πρέπει να περιμένουμε ε, να κάνουμε κάτι εκ των υστέρων. Ε, ε, και ήταν αυτή η σημαντική έκθεση πρωτοβουλίας της, ε, της διαμεσολαβήτριας και θα περιμένουμε να δούμε κατά πώ θα υποβληθούν ε, οι, κάποιες τροπολογίες ή όχι. Γιατί υπάρχουν ε, ε, θέματα στα οποία περιμένουμε να δούμε τι θα πει η Επιτροπή. Κυρίως με το θέμα της διαφάνειας. Εδώ θα πρέπει να προχωρήσουμε γιατί ο μεγάλος αυτός αριθμός των ομάδων εμπειρογνωμόνων που τελικά δεν, ε, δεν συνοψίζονται πουθενά και τον οποίων την ύπαρξη αγνοούμε, ε, νομίζω είναι προβληματικό. Και θα έλεγα, εάν δεν το κάνει η Επιτροπή, και περιμένει μέχρι ότου ολοκληρώσει την έκθεσή της η Επιτροπή για να υπάρξουν ε, ξεκάθαρες ε, οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ για την γνωμοδότηση, θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ε, προσέξουμε να καλυφθεί ολόκληρο το φάσμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Τρούπελ, κυρία Γκρέσλε, αξιότιμα μέλη, είμαι εδώ, είμαι στη διάθεσή σας για να σας ε, ενημερώσω για τις ε, τεχνικές προετοιμασίες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όντως προετοιμάζονται νέοι οριζόντιοι ε, κανόνες για, τους, για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο ακόμα της προετοιμασίας για, την, το πρόγραμμα της οθέτηση τη απόφαση αυτή ε, θα εξαρτηθεί από την πολιτική απόφαση που θα ληφθεί. Δεν μπορώ να σα δώσω άλλε λεπτομέρειε σχετικά. Αλλά όντω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει σύντομα να υιοθετήσει αυτούς τους τεχνικούς κανόνες. Ε, να απαντήσω, Πρόεδρε, ε, στα ουσιώδη θέματα της ε, εισηγήτριας τη κυρία Τρίπελ. Αυτή η συζήτηση όντω ε, γίνεται σε μια πολύ επίκαιρη στιγμή. Ε, θα θυμάστε ότι, η Ευρωπαϊκή, ε, ότι ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στην επιστολή και σε προτάσει ήδη από πέρσι που είχαν υποβληθεί από την διαμεσολαβήτρια και στα πλαίσια αυτά τη απαντήσή του ο κύριο Τίμερμανς έδωσε πολύ λεπτομερεί απαντήσει και ανέλαβε δεσμεύσει τι οποίε τώρα εφαρμόζει η Κομισιόν στα πλαίσια τη αναθεώρησης των οριζόντιων κανόνων τη πολύ σύντομα, αν μπορώ, να μιλήσω για το τι σχεδιάζει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά από όσα προετοιμάζεται να κάνει έχουν να κάνουν με την διαφάνεια, με τη βελτίωση και την αύξηση της διαφάνειας. Να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξεκινούν όλα με τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες εμπρογνωμόνων στο μέλλον θα επιλέγονται, θα στελεχώνονται και θα δημιουργούνται. Έχουμε ένα σύστημα προς το παρόν, σύμφωνα με το οποίο ε, υπάρχουν ε, ε, προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα κράτη-μέλη και θα μέλη κομμάτι ενός διαγωνισμού, αλλά θα μπορούσαν μόνο προς το παρόν. Στο μέλλον θα είναι υποχρεωτικό αυτό. Ε, Βεβαίω αυτό με εξαίρεση των, ε, τους εμπρογνώμονες των δημοσίων αρχών των κρατών μελών. Αυτοί οι διαγωνισμοί θα πρέπει να είναι δημόσιοι. Και αυτό θα γίνεται μέσω ενός νέου μητρώου ε, ομάδων εμπειρογνωμών. Δεν θα είναι δηλαδή κάπου σε μια ιστοσελίδα μια γενική διεύθυνση. Αυτοί οι διαγωνισμοί θα είναι ε, δημόσιοι και θα γίνονται μέσω του νέου Μητρώου ε, για τι ομάδε εμπειρογνωμών. Με αυτό βεβαίω έρχεται και άλλη μία βελτίωση στο σύστημα. Ότι το θέμα τη ισορροπία λύνεται μέσω αυτών των ανοιχτών διαγωνισμών. Οι γενικέ διευθύνσει θα ορίζουν σαφέστατα στου διαγωνισμού του τι προφίλ εμπειρογνώμων να ζητούν. Θα είναι λοιπόν σαφές από την αρχή για όποιον ενδιαφέρεται πώς θα στελεχώνονται αυτές οι ομάδες στο μέλλον. Και μετά, για όποιον ενδιαφέρεται, θα είναι πολύ πιο απλό και θα είναι πολύ πιο προσβάσιμο να δηλώσει το ενδιαφέρον του για να γίνει μέλος αυτής της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Οπότε το θέμα της ισορροπίας θα αποτελεί πολύ μικρότερο πρόβλημα πλέον. Δεν θα είναι κάτι που θα γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Κάτι άλλο που σχετίζεται με τη διαφάνεια πάλι είναι το ότι στο μέλλον θα έχουμε μία, έναν υποχρεωτικό σύνδεσμο μεταξύ των ομάδων των εμπειρογνωμένων που θα εκπροσωπούν κοινά συμφέροντα οι οργανισμούς θα πρέπει να αναφέρονται, να καταγράφονται, να καταχωρούνται στο μητρό των, των ε, λομπιστών. Ε, για να μπορούν να συμμετέχουν να, στις ομάδες τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε στο μέλλον, όταν θα πηγαίνει κανείς στο μητρό αυτών των ε, ομάδων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να υπάρχει ε, σύνδεσμος που θα οδηγεί στο μητρό διαφάνειας. Επίσης, έχουμε ενισχυμένους κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων και για τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων. Στο μέλλον, τα μέλη που θέλουν να εργαστούν σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ως ε, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία αξιολόγησης σύγκρουσης συμφερόντων. Για να γίνει αυτό οι γενικές διευθύνσεις θα έχουν ένα συγκεκριμένο template στάνταρ, πρότυπο, με συγκεκριμένες ερωτήσεις, ίδιες για όλους, τις οποίες θα πρέπει να απαντήσουν οι υποψήφοι. Οι Γενική Διευθύνσεις μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα κάνει την αξιολόγηση του, α, της, της υπόθεσης. Και μετά στο τέλος θα μπορεί κανείς να αποφασίσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, αν, αυτή, αν υπάρχει θέμα σύγκρουση συμφερόντων και αν τελικά ο υποψήφιο μπορεί να είναι μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Αυτά θα καταγράφονται επίσης στο μητρό των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Αυτό αυξάνει συνολικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Επίσης, αναφέρατε την ε, μελέτη που έγινε να κάνω μια αναφορά και εγώ. Όταν δημοσιεύτηκε η μελέτη αυτή, είχε ξεπεραστεί από διάφορες εξελίξεις ε, όπως αυτές που σας ανέφερα. Οπότε η μελέτη αυτή ε, ασκούσε κριτική για διάφορα σημεία. Ε, εν τω μεταξύ όμως η Κομισιόν ήδη δημοσίω είχε α, δεσμευθεί να διαχειριστεί, να διεκπαιρεώσει κάποια από αυτά τα σημεία. τα οποία θεωρούνται ως ε, ε μη επιτυχή. Αυτό ήταν ε, καλό γιατί εκείνη τη στιγμή είχαν γίνει ανακοινώσεις μόνο, τώρα έχουμε περάσει τη φάση της εφαρμογής, αλλά η μελέτη είναι ανακριβής σε πολύ σημαντικά σημεία. Θα μπορούσα να σας δώσω πολλά παραδείγματα, αλλά θέλω να πω το εξή και να το καταστήσω απόλυτα σαφές. Η μελέτη λέει ότι υπάρχουν ανισορροπίες. Καταρχάς, είναι ε, άτυπες αυτές οι πληροφορίες και πολύ γενικόλογες να κάνω ένα σημαντικό σχόλιο για το θέμα της ισορροπίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει μια έτσι ε, διαφοροποιημένη προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει μια ε, ισότητα 50-50 αυστηρά μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων στις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφώς υπέρ, αναφαντών υπέρ της αρχής της ισορροπίας και αυτό το καθιστούμε απόλυτα σαφέ στους κανόνε που θα δημοσιευθούν σε λίγε εβδομάδε, τους νέους κανόνες αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας βαθμός ευελιξίας που να λαμβάνει υπόψη τα συγκεκριμένα καθήκοντα, τη συγκεκριμένη εντολή που θα έχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Μπορεί να έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που να χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα προφίλ και να καταλήξουμε τελικά σε μια σύνθεση που δεν είναι 50-50 αυστηρά και οπωσδήποτε μοιρασμένη. Ε, δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι, αυτό είναι συστημικό πρόβλημα. Ε, η προσοχή μας ε, επίσης ε, δόθηκε και σε διάφορες περιπτώσεις ανισορροπίας και είπαμε ότι θα μπορούσαμε ίσως να τις δούμε μεμονωμένα, αλλά όταν τις μελετήσαμε καλύτερα είδαμε ότι ήταν ανακριβείς οι πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μελετά μια πρόταση και θα την δημοσιεύσει έτσι ώστε να βελτιωθεί συνολικά η λογοδοσία, η νομιμοποίηση, η διαφάνεια σε σημαντικό βαθμό. Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε όλη αυτή τη συζήτηση ή να κάνουμε πιο λεπτομερή ανταλλαγή ε, απόψεων, βεβαίω, Πρόεδρε, είμαστε στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι η διαφάνεια είναι καλό ρυθμιστή τη κατάσταση και μπορεί να ε, προλάβει κάποιε συγκρούσει συμφερόντων. Η κυρία Τρούπελ για να ολοκληρώσει. Ναι, ευχαριστώ. Ε, κοιτάζω τι τροπολογίε των συναδέλφων και θα ήθελα να απαντήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ναι, θα αξιολογήσουμε πολύ προσεκτικά τι προτείνεται, αν επαρκεί ή όχι. Προσωπικά να σας πω ότι όσον αφορά την ισορροπία και το τι σημαίνει για την κοινωνία να εκπροσωπείται στις ομάδες εμπειρογνωμόνων, έχω άλλη άποψη. Αλλά αυτό το οποίο είναι σαφές ε, στην Επιτροπή μας είναι ότι θα είμαστε δίκαιοι, αλλά θα ε, είμαστε και επικριτικοί. Θα δούμε τι θα προτείνετε και αν δεν αρκεί, νομίζω ότι είναι σαφές τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα και έχουμε και τη δυνατότητα να ε, θέσουμε επιφύλαξη. Θα δούμε και ελπίζουμε να μας κάνετε καλές μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ κυρία Τρούπελ. Για τις ε, τροπολογίες, λοιπόν, αν επιθυμείτε να υποβάλλετε τροπολογίες, 8 Μαρτίου 12 η ώρα ε, η λίγη προθεσμία. Θα τις εξετάσουμε και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στι 16 στις 17 Μαρτίου. Η έκθεση θα εξεταστεί στις 23 Μαρτίου και για την... Ε, συγγνώμη, 23 Μαρτίου είναι στην Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού Στις 7 Απριλίου θα εγκρίνουμε το τελικό κείμενο στην Επιτροπή Προπολογισμών και κατόπιν η διαδικασία θα προχωρήσει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Je voudrais vous inviter d'abord... Καταρχάς, ε, βάλτε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες ε, στη συσκευή, να κάνουμε μια επαλήθευση. 34 θα πρέπει να ψηφίσουν. Ψηφίστε παρακαλώ για να ελέγξουμε ότι λειτουργεί καλά. 25, 26, 29, 30... Un c'est bon. Εντάξει. Πρώτη μας ψηφοφορία η έκθεση του συναδέλφου Ντεσόφσκι για την ε, κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την ε, Ενώνα Μουργκλάς στο Βέλγιο. Υπάρχει μια συμβαστική τροπολογία Α. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας. Ευχαριστώ. Ε, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, τροπολογία 9 καλύπτεται από τη συμβαστική α που υπερψηφίσαμε, τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Για το σύνολο της γνωμοδότησης ε, με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται 29 ψήφοι υπέρ, 6 κατά Συγχαρητήρια στο συντάκτη. Τώρα, ψηφίζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για το προσχέδιο προπολογισμού του 2017, τμήμα 3. Εδώ έχουμε διάφορες συμβαστικές προτάσεις. Τροπολογία 1, υπέρ. Πολύ καλή τροπολογία. Κατά. Έτσι λέει ο κύριο Όλμπριχτ και επιβεβαιώνεται. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπερθών 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 26 υποσύρεται 29 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική 7 εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Συγγνώμη. Θα την ψηφίσουμε σε τρία τμήματα για τις ε, τροπολογίες 43, 46 και 47. Το κομμάτι που καλύπτει αυτό... Α, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτο τμήμα. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 σε τέσσερα τμήματα. Για το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Ε, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Να κάνουμε μια επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 10. Πέραση της ψηφοφορίας. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ έναντι 17 κατά. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Επαλήθευση με ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται πάλι 18 ψήφοι υπέρ 17 κατά. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 8. Σε δύο τμήματα. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Έπρεπε να γυρίσω τη σελίδα από την άλλη. Θα ζητώ συγγνώμη. Τροπολογία υπαριθμών 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική 3 εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική 12 εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συμβαστική τροπολογία υπεριθμών 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 15. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία, ε, τροπολογία 112, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές. Θα κάνουμε μια επαλήθευση γιατί δεν είδα όλους να ψηφίζουν. Για την 112 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 16 ψήφοι υπέρ, 17 κατά και 2 αποχές. Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18. Συμβαστική τροπολογία 18, λοιπόν. Υπέρ της συμβαστικής. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 118. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται 18 προς 17 τροπολογία 120, και 126 και 129 που έχουν το δύο αντικείμενο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία υπερψηφίζεται 18 προς 15 μία εποχή. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία γκρίνεται 18 προς 16 μια εποχή. 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ. Είπα 25, συμβαστική υπέρ, κατά. Θα επαληθεύσουμε με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 28 ψήφι υπέρ, 6 κατά μια αποχή. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 186 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 29 με προφορική τροπολογία αλλά χωρίς ε, αυξήσεις φόρων αντικαθίσταται από το φορολογικό βάρος για όλους τους πολίτες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. το σύνολο του κειμένου, για το σύνολο του κειμένου, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Η έκθεση εγκρίνεται 25 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. τον, ο κύριος Στέκοφσκι αντικαθιστά τον κύριο Φερναντές. Για την ε, μεταφορα ένα, 1-2016. Είναι αυτό. Ε, του Δεκεμβρίου 2006 κανονικά ήταν έναν ο Φερνάντες και θα μιλήσω. Monsieur Setkovski, Θα αντικαταστήσατε τον ε, κύριο Φερναντές. Θα αναφερθείτε στο σχέδιο μεταφοράς 1 ε, για τον Ιανουάριο του 2016 Ah, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Μιλούμε για την πρώτη μεταφορά του τρέχοντος έτους από το 4002 το αποθεματικό στο 0004 για το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης το ποσό είναι 1.095.544 ευρώ και αυτό το ποσό θα πάει για υποστήριξη παλαιών υπαλλήλων ε, της βιομηχανίας ε, γυαλιού στην Ευρώπη λόγω της ε, παγκοσμιοποίησης ε, και των ε, συνεπειών που είχε αυτή στον, ε, στον κατασκευαστικό αυτοκλάδο. Άρα πρόκειται μια μεταφορά συνεπής γιατί έχει εγκριθεί προηγουμένως η έκθεσή σας για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Voulez-vous remettre votre carte dans le... <laughs> Bon, est-ce que tu as éclos là Πέρας της Le rapport est adopté. Εγκρίνεται η, η έκθεση 18 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Δεν υπάρχουν, άλλα, α, δεν υπάρχουν άλλες αιτήσει μεταφοράς. Ε, η επόμενη συνεδρία είναι 23 Φεβρουαρίου από τις 3 έως τις 4.30, στις 16 Μαρτίου από τις 9 12.30 και από τις 3 έως τις 6.30 και στις 17 Μαρτίου από 9 12.30.